Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι γιατί θα αρχίσει η συνεδρίαση. Uh, dear colleagues, I would like to start... Παρακαλώ, έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη και ελάχιστο χρόνο για πολύ σημαντικά θέματα, γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Για σήμερα το πρωί θα συνεχίσουμε τη συζήτηση του, της γνωμοδότησης Όλμπριχτ για το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Επίσης, έχουμε και τον ε, αναπληρωτή διευθυντή για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζαν που θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Όλμπριχτ και μετά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Συνέχισε Γιάννη και ελπίζω να ησυχάσουν οι συνάδελφοι. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας δώσω μερικές πληροφορίες για τον τρόπο εργασίας ως προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα τις ε, δημοσιονομικές αρχές, του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Έχουμε συνηθίσει να συζητάμε κυρίως τα ζητήματα των διαρθρωτικών ταμείων. Το πόσα κονδύλια έχουμε δηλαδή και ε, ποια είναι η αποδέκτηση αυτών των κονδυλίων. Αυτό γίνεται με κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό εργασιών, ε, με την προοπτική των, του δημοσιονομικού πλαισίου, των δημοσιονομικών προοπτικών. Το θέμα όμως ε, των δαπανών, του ελέγχου των ε, δημοσιονομικών οργάνων το θέμα των αρμοδιοτήτων των διαφόρων θεσμικών οργάνων στα πλαίσια του προϋπολογισμού και της οικονομίας, όλα αυτά τα θέματα ρυθμίζονται σε άλλα έγγραφα και νομοθετικές πράξεις. Πριν από μερικά χρόνια και πάλι ήταν αρμόδιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα πάλι ασχολούμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το θέμα της αναθεώρησης του εξυγχρονισμού του δημοσιονομικού κανονισμού. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά ένα έγγραφο που κατήρτισε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προκάλεσε σφοδρές συζητήσεις, όχι μόνο στην Επιτροπή αλλά και στο Συμβούλιο, θα ήθελα λοιπόν να γύρω το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό, γιατί είναι πραγματικά συνήθιστα περίπλοκο ζήτημα και όχι και πολύ ελκυστικό. Γιατί αφορά πολύ συγκεκριμένους τεχνικούς κανόνες που αφορούν τις δημοσιονομικές ροές και τον έλεγχο. Η κυρία Γκρέσλα είναι η συγγετρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μαζί με μια ομάδα εργασίας που έχει συστηθεί εδώ και αρκετούς μήνες εκπονεί την εκδοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με νομοθετικό κείμενο, γι' αυτό η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συγκροτηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να, υποβάλει, να περιλαμβάνει τροπολογίες σε αυτό το δημοσιονομικό κανονισμό. Οι τροπολογίες αυτή τη στιγμή είναι αρκετές. Και η συζήτηση που έχει ξεκινήσει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιστρέφεται γύρω από το θέμα του βαθμού ανάλυσης και το πόσο ειδικέ θα είναι οι τροπολογίες που θα υποβάλουμε. Αυτό είναι το γενικό κλίμα της συζήτησης και θα να σας πω ότι τα κράτη-μέλη, δηλαδή το στο Συμβούλιο, θα προτιμούσαν ο κανονισμός είναι όσο γίνεται πιο γενικός. Να μην είναι πολύ ειδικό και α, διεξοδικός. Να μην έχει πολλές τομεακές ρυθμίσεις. Αυτή είναι η γενική ε, προσέγγιση στο Συμβούλιο και αυτό μας το επαναλαμβάνω πολύ συχνά. Να μην ε, γίνει πολύ διεξοδική αναλυτική ρυθμίση για να παραμείνουν οι αρμοδιότητες στους τομεακούς κανονισμού. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάνν. Είναι απαράδεκτο ευρωβουλευτές να μιλούν είτε μεταξύ τους είτε με τους βοηθούς, τους, γιατί πραγματικά έτσι δημιουργείται μια φασαρία στην αίθουσα και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε καθόλου τον εισηγητή. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως διαφορετική από αυτή του Συμβουλίου. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να διαθετηθούν, να ρυθμιστούν, γιατί μπορεί να δοθεί εντύπωση ότι ο τρόπος προσέγγισης του, της ηγήτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι απόλυτα δεκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι εμείς προτείνουμε να περιληφθούν στον κανονισμό κάποιες ρυθμίσεις που είναι υπερβολικά αναλυτικές, υπερβολικά εξειδικευμένες και άπτονται περισσότερο τομεακών ρυθμίσεων. Πολύ συχνά ακούγεται η γνώμη ότι το Κοινοβούλιο ε, θέλει να ασχοληθεί με τη μικροδιαχείριση, το micromanagement. Ότι θέλουμε δηλαδή εμείς όλες τις λεπτομέρειες να τις ρυθμίσουμε ήδη στον κανονισμό. Είναι αναφυσβήτητο ότι Όλη η προσπάθεια της εισηγήτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθεί, ε, όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται να, για να περιλάβει ορισμένα στοιχεία των εκτελεστικών κανονισμών στον δημοσιονομικό κανονισμό. Γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συναποφασίζει αφενός, αλλά ταυτόχρονα να συνελέγχει, να συμμετέχει στον έλεγχο της διεξαγωγής ορισμένων δημοσιονομικών δραστηριοτήτων. Από τη μια πλευρά δηλαδή έχουμε τη θέση της εισηγήτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να υπησέλθει σε πολλές λεπτομέρειες του δημοσιονομικού κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ μιας ε, εξειδίκευσης αλλά όχι μεγάλης, ενώ το Συμβούλιο προτιμά να παραμείνει σε μια γενική διατύπωση και τις λεπτομέρειες του τομεακούς κανονισμούς. Οι εργασίες για το δημοσιονομικό κανονισμό, δηλαδή η νομοθετική διαδικασία, καλό θα ήταν, ε, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. Δηλαδή το θέμα επήγει και απαιτείται να ανασκουμποθούμε και να επιταχύνουμε τις εργασίες μας γιατί το οριστικό κείμενο των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξεταστεί αμέσως μετά τις θερινές διακοπές. Αυτό που προτείνω εγώ είναι ένα μικρό απόσπασμα που αφορά κάποια στοιχεία μόνο του δημοσιονομικού κανονισμού, κυρίως αφορά την επιμερισμένη διαχείριση, το shared management που λέμε. Και αυτό αφορά και την κοινωνική πολιτική και την περιφερειακή πολιτική. Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρω ρητά ότι εφόσον μιλούμε για επιμερισμένη διαχείριση, για το shared management, αυτό προϋποθέτει ότι κάποιες εκτελεστικές ε, δραστηριότητες, εφαρμοστικές, εκχωρούνται στα κράτη-μέλη. Αυτό προβλέπει η τροπολογία υπαριθμών 3. Και νομίζω ότι είναι η διατύπωση αυτή πολύ συγκεκριμένη. Φαίνεται προφανής βέβαια, αλλά καλό είναι να το αναφέρουμε. Γιατί από τη στιγμή που πρόκειται για επιμερισμένη διατύπωση, ορισμένα εκτελεστικά καθήκοντα μεταβιβάζονται στα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια διαθέτησης κάποιων θεμάτων που ήταν πολύ σφοδρά και προκάλεσαν έντονη συζήτηση σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Θα ήθελα συνοπτικά να σας πω ότι η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το θέμα ποιος δικαιούται να διαπιστεύσει τα Τα τους διαχειριστικούς οργανισμούς ε, που ασχολούνταν με τα διάφορα προγράμματα. Η συγκήτρια του Κοινοβουλίου ε, και το Κοινοβούλιο και το, ε, η Επιτροπή πιστεύουν ότι σε κάθε κράτος μέρος θα πρέπει να υπάρχει ένας μία αρχή διαπίστευσης που να είναι αρμόδια για τη διαπίστευση των οργανισμών και επίσης είναι αρμόδια η Επιτροπή αυτή τα διαπιστευμένα όργανα να ελέγξει αν όντως εκτελούν τα καθήκοντά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη συζήτηση εξετάστηκε μήπως θα έπρεπε ε, η αρχή της διαπίστευσης ε, να αναχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι αρμόδια για τη διαπίστευση όλων των διαπιστευμένων οργανισμών, αυτών που διαχειρίζονται δηλαδή τα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτό το θέμα ανέκυψε. Η διαδικασία διαπίστευσης είναι πολύ χρονοβόρα όμως και ίσως δημιουργήσει προσκόμματα στην εύρυθμη εκτέλεση των προγραμμάτων. Μέχρι στιγμή πάντω προτείνονται οι αρχέ διαπίστευση να βρίσκονται σε επίπεδο κρατών μελών. Οπότε τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν μεγάλο τμήμα τη αρμοδιότητα για την εφαρμογή τη πολιτική. Η αρχή διαπίστευση προβαίνει στη διαπίστευση συγκεκριμένων οργανισμών, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των επιχειρησιακών των λειτουργικών προγραμμάτων. Τώρα, ποιοι οργανισμοί θα λάβουν διαπίστευση, αυτό εξαρτάται από την αρχή διαπίστευση ενό κράτου μέλου. Έχουμε δηλαδή δύο όρους, τη διαπίστευση και τον διαπιστευόμενο. Έχουμε την αρχή διαπίστευσης και τους διαπιστευμένους οργανισμούς. Αν κοιτάξετε την τροπολογία 5, θα δείτε την πρότασή μου για την αρχή διαπίστευσης. Εκεί αναφέρεται ότι η αρχή διαπίστευσης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των διαπιστευμένων οργανισμών με τα κριτήρια διαπίστευσης. Διακόπτει ο μιλήτης. Επαναλαμβάνω λοιπόν στην τροπολογία 5 έχετε τις πληροφορίες και για τις αρμοδιότητες των διαπιστευμένων οργανισμών. Βλέπετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Στον κανονισμό περιλαμβάνονται και κάποιες πληροφορίες για την ευθύνη και των διαπιστευμένων οργανισμών που υποχρεούνται να υποβάλουν ετήσια καθάριση λογαριασμών. Και αυτό προβλέπεται να γίνει μέχρι την 1η Μαρτίου του επόμενου διαχειριστικού έτους, του επόμενου οικονομικού έτους. Και το αναφέρω αυτό γιατί και στη δική μας Επιτροπή συνεχίζονται ακόμη οι συζητήσεις για το πώς ε, διεξάγεται η διαδικασία της απαλλαγής. Πολύ συχνά η Επιτροπή ε, εξετάζει το θέμα της δυνατότητας επιτάχυνσης της διαδικασίας της απαλλαγής. Από αυτό τον κανονισμό προκύπτει ε, αδυναμία επιτάχυνσης της απαλλαγής, γιατί η απαλλαγή πρέπει να γίνει μετά την έλευση του συγκεκριμένου έτους. Εδώ υπάρχει η συγκεκριμένη πληροφορία ότι μέχρι την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους θα πρέπει να παραχθούν στην Επιτροπή τα στοιχεία για την εκαθάριση των λογαριασμών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για τη συζήτηση των ε, διαρθρωτικών ταμείων και των ευρωπαϊκών ταμείων. Υπάρχει το θέμα της ε, δήλωσης διαχείρισης, ε, διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας. Με βάση την δήλωση αυτή που την υποβάλλει ο διαπιστευμένος οργανισμός, δηλαδή ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του λειτουργικού προγράμματος, έχει και την ευθύνη να υποβάλει αυτήν την ε, δήλωση διαχείρισης, Management Declaration. Και συνεχίζεται ακόμη η συζήτηση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας. Συνεχίζεται, επαναλαμβάνω, αυτή η συζήτηση και από ό,τι φαίνεται δεν θα ευοδοθεί και με επιτυχία. Γιατί δεν θα είναι τελικά υποχρεωτικές αυτές οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Στον κανονισμό αυτό θεσπίζεται η υποχρέωση των διαπιστευμένων οργανισμών να υποβάλουν τις δηλώσεις διαχείρισης. Στην δική μου γνωμοδότηση βλέπετε ποιες είναι οι ευθύνες αφενός της αρχής διαπίστευσης και αφετέρου των διαπιστευμένων οργανισμών. Και επίσης ε, φέρονται και οι ευθύνε και υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με επιμερισμένη διαχείριση, shared management, για μας, τον κανονισμό μας ε, και για την πολιτική συνοχή, όταν ε, μιλάμε για πολιτική συνοχή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν μία αρχή διαπίστευσης και επίσης αυτή η αρχή διαπίστευσης θα είναι αρμόδια για τη διαπίστευση κάποιων οργανισμών. Ένα άλλο στοιχείο που εμφανίζεται στον κανονισμό είναι και το θέμα των σφαλμάτων και κυρίως ε, το θέμα του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος. Και αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη συζήτηση βέβαια. αλλά έχει θέμα, έχει σχέση με την ε, πολιτική συνοχή, γι' αυτό και με αφορά άμεσα. Γίνεται λόγο λοιπόν για το αποδεκτό κίνδυνο σφάλματο. Το ελεκτικό συνέδριο, για παράδειγμα, θεωρεί ότι το αποδεκτό ποσοστό σφάλματος ε, ε, στην πολιτική συνοχή θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο υψηλό. Τι, γίνεται όμως σε περίπτωση που είναι τόσο υψηλό το σφάλμα. Βέβαια, άλλο επίπεδο σφάλματος και άλλο επίπεδο παρατυπιών. Το επίπεδο σφάλματος είναι κυρίως ο κίνδυνος σφάλματος. Και υπάρχει και το θέμα του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος. Στον κανονισμό αυτό υπάρχει μια πρόταση να περιλάβουμε και την έννοια του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος. Έτσι αποκλείονται όμως ε, ορισμένες ε, δραστηριότητες. Θα πρέπει, ε, αναφέρομαι λοιπόν, κάποιες δραστηριότητες που ε, περιλαμβάνουν ένα πολύ ψηλό κίνδυνο σφάλματος δεν θα πρέπει να αναλαμβάνονται. Αυτό όμως προϋποθέτει μια εξάντε, μια εκ των προτέρων αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων. Το ελεκτικό συνέδριο χρησιμοποιεί κάποιες ε, διεθνείς ε, Προδιαγραφέ για τον κίνδυνο σφάλματο και χρησιμοποιώ αποδεκτό ποσοστό σφάλματος το 2%. Αυτό είναι το μέτρο που χρησιμοποιεί το ελεγκτικό συνέδριο. Το θέμα είναι για τις καινοτόμες δράσεις της ε, πολιτικής συνοχής μπορούμε να αποδεχτούμε ένα υψηλότερο ποσοστό κίνδυνο σφάλματος ή όχι. Ανακεφαλώνοντα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι καταρχήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με το δημοσιονομικό κανονισμό που είναι νομοθετικό κείμενο. Στο κείμενο αυτό υπάρχουν κάποια αποσπάσματα που αφορούν όλες τις πολιτικές. Υπάρχει ένα τμήμα που άπτεται της επιμερισμένης διαχείρισης. Στην γνωμοδότηση που καταρτίζω εγώ για την Επιτροπή μας, επικεντρώνομαι στο θέμα της επιμερισμένης διαχείρισης, που περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εφαρμογή τη πολιτική συνοχή. Αφορούν αφενός τη διαπίστευση και αφετέρου τον περιορισμό των ε, οργανισμών. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τις, ε, τους διαχειριστικούς οργανισμούς, τους φορείς πληρωμής και τις αρχές διαπίστευσης. Έχουμε πολλούς οργανισμούς και φορείς. Η συγκεκριμένη πρόταση προτείνει την διαπίστευση να την εξασφαλίζουν οι διαχειριστικοί οργανισμοί. Αντί για τρεις οργανισμούς σε κάθε χώρα, σε τρεις ε, σε κάθε χώρα να έχουμε δύο φορείς, δύο οργανισμούς. Νομίζω ότι έτσι απλουστεύουμε κατά πολύ τη διαδικασία, περιορίζοντας από τρεις τους φορείς σε δύο. Σας ευχαριστώ, Γιάννη. δημοσιονομική αρχή, για τις δημοσιονομικές αρχές. Όσο η δημοσιονομική αρχή α, δείχνει και υπογραμμίζει την διαχείριση σε επίπεδο μικροοικονομικών του προπολογισμού, τόσο η ίδια δημοσιονομική αρχή επομίζεται επιχειρησιακές ευθύνες εντός αγωγικών. Επομίζεται. Και αυτό επικρίνεται και από τους φορείς ελέγχου για λόγους διαχείρισης και για λόγους διαχωρισμού καθηκόντων μεταξύ εκείνων που ε, θεσμοθετούν, θεσπίζουν νομοθεσία και εκείνων που εκτελούν, χρειάζεται ένα καλό σύνορο, μια καλή διαχωριστική γραμμή όσον αφορά τις ε, ευθύνες. Και αυτό είναι αναγκαίο για να πετύχουμε το στόχο της απλούστευσης. Απλούστευσης όσον αφορά την εφαρμογή του κειμένου. Ξέρετε ότι είναι ένα στόχος επί το οποίου 23 υπουργοί έστειλαν αποστολή στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον επίτροπο υπεύθυνο για θέματα προπολογισμού ε, για να εκφράσουν τι ε, προσδοκίε του. Είναι και δική μα προσδοκία. Και μέσω του διαλόγου με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο θα θέλαμε να επιφέρουμε αυτή την απλούστευση που στο κάτω-κάτω θα εξυπηρετεί του δικαιούχου. Θα μπορούν να λαμβάνουν και χειρίζονται αποτελεσματικότερα τα κοινοτικά χρήματα. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση που ετοίμασε και ο Σάμπριτ και την πρόταση που κάνει, τη που κάνει, έχω δύο-τρία σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, θα έλεγα ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι εν γέννη με την πρόταση του κ. Έχω δύο πράγματα να πω. Όσον αφορά το θέμα τη επενδυσμένη διαχείριση άρθρο 56 του σχεδίου κανονισμού των αθεωρημένων, έχουμε δύο τροπολογίες οι οποίες μας δημιουργούν πρόβλημα. Αυτές είναι η τροπολογία 4, η οποία υποχρεώνει να αντικατασταθεί ο όρος ε, δύναται με το, το may με σάλ ότι πρέπει, ότι θα, σάλ γίνεται υποχρεωτικό. Η Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε, ε, έχω φτάσει στα όρια μου. Θέλω να ζητήσω του πολιτικού συμβούλου και του βοηθού να φύγουν από την αίθουσα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Καταλαβαίνω ότι σα ενδιαφέρουν πολύ τα επόμενα σημεία. Είμαστε στο πρώτο σημείο ε, τη ημερήσια διάταξη και κάνετε δύνατη τη δουλειά μα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ε, και ο Πάτρο Καλέτα. Σας παρακαλώ, θέλουμε τα μέλη τη επιτροπή θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μα και εσεί δεν μα αφήνετε να δουλέψουμε. Το κάνετε αδύνατο. Και λυπάμαι, αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση. Εάν συνεχιστεί η κατάσταση, θα ζητήσω όλοι οι βοηθοί να αποχωρήσουν από την ε, αίθουσα. Συγγνώμη, συνεχίστε κύριε. Ευχαριστώ. Ε, καταρχάς λοιπόν την τροπολογία 4 που προτείνει ο κ. Σόλμπρεκτ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί υποχρεωτικά όλα τα συστήματα διαχείριση και ελέγχου των καταμελών υποχρέωση που συνεπάγεται την χρήση μέσων που δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εάν θεωρήσουμε ότι θα ήταν καλό να προχωρήσουμε σε ελέγχους, επιχειρήσεις ελέγχου, σποραδικούς ελέγχους να κάνουμε στα κάτι μέλη, εντάξει, αλλά γενικά να διεξάγονται οι έλεγχοι με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι κάτι που μας δημιουργεί ένα πρόβλημα διαχείρισης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό θα δημιουργούσε και μεγάλους κινδύνους καθυστερήσεων για την έναρξη των προγραμμάτων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει το δύνατε ΜΕΙ που μας αφήνει ένα περιθώριο ευελιξίας. Άλλη ανησυχία που έχουμε στον αφορά τροπολογίες του κ. Όλμπερτ αφορά την τροπολογία 3 η οποία καταργεί την υπόθεση των 100 μελών επιβάλλουν κυρώσεις στους δικαιούχους εφαρμόζοντας το ευρωπαϊκό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο και αυτή η διαγραφή θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητη. θα θέλαμε λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι αυτή που θα ληφθεί υπόψη, αυτή που θα ισχύει αν προφανώς συμφωνεί ο κύριος εισηγητής και αν συμφωνεί και η Επιτροπή σας όσον αφορά τον ανεκτό, τον ανεκτό κίνδυνο σφάλματος όπως είπε και ο Σάλμπερτ είναι εξειδικευμένο περιπλοκότατο ζήτημα το ελεγκτικό συνέδριο έκανε κάποιες προτάσεις στην πρόσφατη έκθεσή του ζήτησε να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτού του κινδύνου σφάλματος που θα μπορούσε να είναι ανεκτός πέραν του οποίου για να προστευτούν τα πράγματα το κόστος του ελέγχου είναι τέτοιο που είναι μεγαλύτερο από την πιθανότητα εξοικονομήσεως ποσών, άρα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Δεν λέμε να μειώσουμε τους ελέγχους, θέλουμε να φροντίσουμε ούτως ώστε η έλεγχη είναι ανάλογη, αναλογική. γίνεται μεγάλη συζήτηση στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη και το ελεκτικό συνέδριο που έκανε αρχικά αυτή την πρόταση προβάλλω μια αντίσταση, στεναρή αντίσταση. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη και το ελεκτικό συνέδριο σε αυτή την πρόταση. Πρότασή του είναι να αξιολογεί τον κίνδυνο σφάλματο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι και αυτό να μην προβλέπεται στο νομοθετικό κείμενο, αλλά στα έγγραφα που θα είναι προσαρτημένα στι τομεακέ προτάσει ε, των δημοσιονομικών δελτίων που, που διατίθεται στη ε, νομοθετική αρχή. Αυτή είναι η λύση. Αυτή Έτσι τροποποίησαμε, έτσι αλλάξαμε αυτή τη δική μας πρόταση όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μισό λεπτό ακούστε τι έχω να σα πω. Να σα προτείνω το εξή. Γιάν, και σε σένα απευθύνομαι. Να διακόψουμε τη συζήτηση αυτού του σημείου τη μερική διάταξης και να ψηφίσουμε διότι η συνέχιση της συζητήσεως υπό αυτές τις συνθήκες είναι δυσχερέστατη. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση αφού κάνουμε τις ψηφοφορίες. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ακούσαμε τις απαντήσεις, εξηγήσει που χρειάζονται. Εάν θα είχα την καλοσύνη να πείσετε ένας από τους συνεργάτες σας μαζί μας, γιατί να συνεχίσουμε μετά την ψηφοφορία, θα το εκτιμούσαμε αν το κάνατε αυτό, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κάνουμε αυτό που πρότεινα. Να διακόψουμε δηλαδή τη συζήτηση. Συμφωνείτε. Ιαν. συμφωνεί. ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τώρα τις ε, ψηφοφορίες. Uh, right our not members, and we, we will do a check. Do The machine will tell us, but also that the members they want to have. Okay. Uh, dear, dear colleagues, in particular, dear... Συνάδελφοι, αγαπητοί συντονιστέ, όλου ιδιαίτερου, σα παρακαλώ, κάντε έναν έλεγχο, κοιτάξτε αν τα στατεύματά σα είναι στην αίθουσα. και θα δούμε και στι οθόνε. θα κάνουμε έναν έλεγχο αν δεν ψηφί, να μην ψηφίσουν παραπάνω από αυτοί που πρέπει αλλά πρέπει να δείτε κατά πόσο είστε αυτοί που πρέπει στον αριθμό. Ας κάνουμε και ένα ηλεκτρονικό έλεγχο να δούμε αν δουλεύουν οι κάρτες σας. Σας παρακαλώ λοιπόν βάλτε την κάρτα σας στο μηχάνημα για να κάνουμε τον έλεγχο. Λοιπόν, έναρξη της δοκιμής, της δοκιμαστικής πληροφορίας. Uh, yeah. Έχουμε πέντε μέλη του ΕΛΚ παραπάνω, αλλά και σοσιαλιστές. Είναι ένας σοσιαλιστής πιο παραπάνω. Ένας σοσιαλιστής. No, it's okay. Όχι, εντάξει. Γιούτα. Γιούτα είμαστε εντάξει τώρα. Okay, dear colleagues, we, are now okay with socialists. Λοιπόν, εντάξει, οι σοσιαλιστές, έχουμε έναν παραπάνω στο ΕΛΚ. And just, we, we are following. We, we, we re restart. We open again. Can we, can we restart? Λοιπόν, ας ξανακάνουμε τον έλεγχο αν θέλετε. Ξανακάνουμε τον έλεγχο για να είμαστε σίγουροι. Uh, open, λοιπόν, ξεκινά η δοκιμαστική ψηφοφορία. Εντάξει, μπορείτε ακόμα να ψηφίσετε. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω.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 θα με διορθώσει ο Πίπερ αν κάνω λάθος, είχαν 569 τροπολογίες και περίπου 30 συμβαστικές συντάξαμε με μετά από διαπραγματεύσεις. 30 τροπολογίες συμβαστικές. Θα θυμόσαστε ίσως ότι και η Επιτροπή Απασχόληση ανακατεύθηκε μέσω του άρθρου 50 στην ετοιμασία αυτής της εκθέσεως και οι προτάσεις της νομοδοτήσεως της Επιτροπής Απασχολήσεως θα υθετηθούν άνευ ψήφου διότι εκεί που έχουν αρμοδιότητα αυτοί αποφασίζουν. Εκεί που δεν έχουν θα ψηφίσουμε στις τροπολογίες. Νομίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα. Ξεκινάμε λοιπόν από την τροπολογία 59 υπέρ κατά απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 61 ξεκινάει τώρα ο έλεγχος EPP. E Έχουμε δύο μέλη του ΕΛΚ πάνω από το όριο. Πρέπει λοιπόν να επαναλάβουμε τη ψηφοφορία. Παρακαλώ τους συναδέλφους του ΕΛΚ να προσέξουν. So we open the vote. Επανάληψη λοιπόν της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. E Ένα μέλος του ΕΛΚ. Sorry. So we open again. We'll see if the machine tells us if someone takes out, who takes out. Could somebody take out maybe disappear? No. It's not. So we have to again reopen the vote. Με επανάσταση ψηφοφορία. We open the vote. Yeah, we open the vote. Έναρξη ψηφοφορία. Well, again, EPP, one person. Ξανά έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ θα αφαιρέσουμε μία ψήφο. Το ΕΛΚ είναι κατά, από ό,τι ξέρω. Ξανά, λέει η γραμματεία, επανάληψη της ψηφοφορίας. It's fine. It's fine now. Okay. So of course we close. <laughs> We close We Λοιπόν, πέρας. 24 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 65 έχουν προφορική τροπολογία αν δεν είναι κανείς εναντίον της προφορικής τροπολογίας και δεν έχουμε κάποιον κατά ψηφίστε τροποποιηθεί τροποποιήθη 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 66 κατά 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ μάλιστα κύριε Πίπερ στην λίστα ψηφοφορία υπάρχει ένα σφάλμα. Εγώ θα συστήσω ω Λαϊκό Κόμμα να υπερψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Ε, εννοείται την 72. Α, 73, 73. Ναι, Λαμπέρ. Ψηφίσαμε ήδη την 72. Α, ωραία, τότε είναι σαφέ. 73 λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, ο εισηγητή είναι θετικό για την 73 και πρόκειται για τον αθλητισμό, έτσι δεν είναι. Εμένα μου αρέσει ο αθλητισμός. Λοιπόν, το Λαϊκό Κόμμα το υποστηρίζει. Υπέρ λοιπόν του 73, κατά, αποχές εγκρίνεται, 74 αποσύρεται, συμβιβαστική ένα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα πάμε στην 75 δεύτερο μέρος. Μόνο το δεύτερο μέρος θα ψηφίσουμε τις 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100. Όχι. Α, εκπίπτει αυτή καλώς. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν δεκαεννέα υπέρ. Κατά υπέρ λοιπόν ακόμα κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 120 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, την 120 πάντοτε, έναρξη ψηφοφορίας. Δύο ψήφοι του Λαϊκού Κόμματος είναι άνω του ορίου, δύο υπερβάλλουσες. Τώρα μία, λέει η Πρόεδρος, μία παραπάνω. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία και πάλι, ε, για την 120. Πέρας. Εγκρίνεται 24 υπέρ 21 κατά. 121 με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κανείς που είναι αντίθετος με την προφορική τροπολογία. Όχι καλά. Λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 122 αρχίζει. Πάλι μία ψήφο παραπάνω του Λαϊκού Κόμματο. Είναι μία παραπάνω, λυπούμε λέει η Πρόεδρος. Είμαστε αναγκασμένοι να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για να μην μας κατηγορήσουν κατόπιν για αταξίες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με, όπως βλέπετε, μία ψήφο διαφορά. Γνωρίζει το Λαϊκό Κόμμα τι κάνει, λοιπόν. 123 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά. Αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Εάν κάποιος από σας φωνάξει επαλήθευση, α, καλά, ωραία, επαληθεύουμε λοιπόν. 125 αρχίζει η ψηφοφορία. πάλι μία ψήφος του Λαϊκού Κόμματος πάνω από το όριο. Ξαναρχίζουμε να αφαιρεθεί μία κάρτα του Λαϊκού Κόμματος. Ξαναρχίζουμε. 125. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική. Ορίστε παρακαλώ να πω στους συναδέλφους μου, όσοι ψήφισαν μόλις τώρα και που είναι ο σωστός αριθμός, αυτοί μόνο να ψηφίζουν και στο μέλλον. Και να μείνουν βεβαίως, να μην φύγουν. Δεν έχω καμία διάθεση απολύτως να παρενοχλεί την ψηφοφορία. Όσοι ψήφισαν, αυτοί να συνεχίσουν να ψηφίζουν. Και η πρόεδρος θα είναι ευχαριστημένη και εγώ. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 Συμβαστική 8, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 171 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. 171. Πάλι μία ψήφος του ΕΛΚ παραπάνω. Λοιπόν πολύ, ξαναρχίζουμε την ψηφοφορία. 171. Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μηχάνημα, λέει ο Πρόεδρος. Ξαναρχίζουμε την ψηφοφορία. 171. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 173 με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει ένσταση κατά αυτής, ψηφίζουμε υπέρ της 173 κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 εκπίπτει 81 was rejected. Rejected.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 Παρακαλώ και οι υπόλοιποι ε, της γραμματείας να παρακολουθούν προσεκτικά ώστε να μπορούμε να αντιδρούμε ταχύτατα. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, θέλετε επαλήθευση. Καλά λοιπόν. Για μένα όμως ήταν σαφές. 184 εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Δεν είναι Μάρκο 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201 μου λέει η συνεργάτη μου υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αυτή θέλετε τσεκ ωραία 201 επαλήθευση αρχίζει πάλι μια ψήφωση του Λαϊκού Κόμματος παραπάνω Βανίστερ Ρόι. Το ποντίκι η γάτα παίζει τώρα, πρέπει να δω. I don't know about, they στο μεταξύ μπορεί κάποιος από τους πολιτικούς συμβούλους να ελέγξει. Το Λαϊκό Κόμμα διαθέτει εδώ 17 μέλη μαζί με την ε, Πρόεδρο. Μήπως δεν με έχετε υπολογίσει εμένα. Ας, ας εγερθούν παρακαλώ τα μέλη του Λαϊκού Κόμματος. Νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολο να σας μετρήσουμε.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

got all the titulars except uh, two. So they have to be It's up to the group to decide uh, who votes. Yes, yes, no problem. Tenemos los, todos los titulares menos dos, ¿no? Estarás y Nicolás. Nicolás y Estarás no está, y estaras No está. Okay. We, we have... Uh, Are we finished? Μήπως τελειώσατε? Can we... Can we resume the vote? Μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία 201. Ηλεκτρονικά 201. Αρχίζει η ψηφοφορία. 201. Αρχίζει. πέρας εγκρίνεται και με μεγάλη διαφορά. Πρέπει να επιστρέψουμε στις 176 και 177. Μετά από έλεγχο προκύπτει ότι πρέπει να τις ε, ψηφίσουμε. 176 υπέρ. Ε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές αυτή απορρίπτεται τώρα ξανά στη 202 υπέρ κατά υπέρ μάλλον συγγνώμη ακόμη υπέρ κατά αποχές χρειάζεται επαλήθευση 202 έναρξη δεν θέλω καν να κοιτάξω την οθόνη για να μην επηρεαστώ πέρας και απερίφθη. 203 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή. 209 υπέρ, κατά αποχές αυτή απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά σε επαληθεύσουμε 208 σύντομη επαλήθευση αρχίζει πέρας απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 εκπίπτει αυτή άρα προχωρούμε στη 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ 215. Υπέρ λοιπόν, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 216. Κατά, αποχές, αν δεν διαμαρτύρεται κανείς. 216 την επαληθεύουμε λοιπόν. Αρχίζει. Πέρας. 24 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Διακόσια είναι δύσκολη η ψηφοφορία. Αν κάποιο διαπιστώσει κάποια ανομαλία να μας το πει αμέσω. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Θα διακόψουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, παρακαλώ εσείς. 218. Uh, it, it fell αυτή εξέπεσε διότι ε, εγκρίθηκε 216. ...225 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... ...226 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... ...227 υπέρ... ...κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα της 228 αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας απερίφθη 229 υπέρ κατά αποχές αυτή νομίζω απορρίπτεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 231 υπέρ κατά θα την ελέγξουμε, θα την επαληθεύσουμε. 231 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 <clears throat> μάλλον και 34 γιατί είναι ταυτόσιμες <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή συμβιβαστική 11 υπέρ κατά Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 253. Ναι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Οι ε, αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. 55 ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 256 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται συμβαστική 12 η κυρία Κρέλ θέλει να λάβει το λόγο παρακαλώ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε νομίζω ότι είναι από τα πιο δύσκολα μέρη της ψηφοφορίας εδώ στην λίστα ψηφοφοριών έχουμε τρεις συμβαστικές τροπολογίες, την 12 του εισηγητού για την παράγραφο 21, την 14 για την παράγραφο 23 και την τροπολογία της δικής μου πολιτικής ομάδας που περιλαμβάνει, αναφέρεται μάλλον και στις δύο παραγράφους. Είναι βέβαια δύσκολη η απόφαση τώρα, αλλά είμαι πεπισμένη ότι εάν ψηφίσουμε χωριστά τις δύο παραγράφους με τις συμβαστικές δηλαδή τροπολογίες του ισίου του μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα αυτό διότι θα παραμείνουν μεμονωμένες παράγραφοι χωριστές. Εμείς έχουμε υποβάλει μια συμβαστική τροπολογία που τη συνδέει και που νομίζουμε ότι κάνει τα πράγματα πολύ σαφέστερα από τις συμβαστικές του του. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πρώτα να ψηφιστεί η τροπολογία 12 της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και μετά οι τροπολογίες 12 και 14 του εισηγητού. Ο κύριος Βανίστερο, όχι. Ωραία. Ε, εγώ θέλω μόνο να πω, λέει πρόεδρος, να σας εξηγήσω πολύ σύντομα. Έχουμε την παράδοση στην Επιτροπή μας ότι δίνουμε στους εισηγητές την δυνατότητα να προτείνουν την σειρά των τροπολογιών για να ψηφιστούν. Τώρα υπάρχει βέβαια η πρόταση αυτή, την οποία υποβάλλει η κυρία Κωνσταντσε Κρέλ, συντονίστρια της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και προτείνω να ψηφίσουμε την σειρά της ψηφοφορίας. Ναι, ναι, ακόμα δεν έχω τελειώσει τη συζήτηση. Ορίστε, ο κύριος Μάρκος Πίπερ. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να λάβω και εγώ το λόγο για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ε, ως εισηγητής μου φαίνεται η σειρά αυτή που έχω προτείνει λογική. Για τις διάφορες κατηγορίες στόχων έχουμε κάνει συμβασμούς, συμβαστικές τροπολογίες δηλαδή, θα τις ψηφίσουμε τώρα. Δεν θα προκαταλάβουμε τίποτα στις ψηφοφορίες αυτές. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε τι στάση θα τηρήσουμε στην ψηφοφορία. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί άραγε να αλλάξουμε την σειρά της ψηφοφορίας, διότι επί της ουσίας, κατά τη γνώμη μου, δεν αλλάζει απολύτως τίποτε, εάν ψηφίσουμε με τον τρόπο που έχω προτείνει. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Γι' αυτό και θα συστήσω να παραμείνουμε στην σειρά που έχει τις τροπολογίες ή λίστα ψηφοφορίας. Η κυρία Σουέντερ. Επισημαίνω ότι στον γύρο διαπραγματεύσεων συζητήθηκε το θέμα αυτό και στην ουσία συμφωνήσαμε όλοι ότι εάν μπορούν οι δύο αυτές τροπολογίες να συγχωνευτούν σε μία, όπως έγινε με την πρόταση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και όλοι συμφώνησαν στον γύρο διαπραγματεύσεων και η γραμματεία είπε ναι. Είπαμε τότε η κοινή τροπολογία για παραγράφους 21 και 23 να ψηφιστεί πρώτη αυτό θεωρήθηκε λοιπόν στο γύρο των διαπραγματεύσεων όπως είπα που κάναμε, που διεξαγάγαμε οι συντονιστέ, ότι θεωρήθηκε σωστό. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ξαναεμφανίζεται στη λίστα ψηφοφορία με διαφορετικό τρόπο. Βανίστελ Έχουμε βέβαια από την συντονίστρια των σοσιαλιστών και με υποστήριξη των πρασίνων ξεκάθαρη πρόταση και βεβαίως και την ξεκάθαρη στάση του εισηγητού, το Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει την ε, θέση του εισηγητού. Όπως είπατε, ας ψηφίσουμε. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπορούμε να επαναλάβουμε τα επιχειρήματα κατέρωθεν, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να προχωρήσουμε την ψηφοφορία. Α, είναι και οι φιλελεύθεροι που ε, θέλουν να λάβουν το λόγο. Εμείς υποστηρίζουμε την θέση του εισηγητού. Είναι σαφής λοιπόν η κατάσταση, υπάρχει διάσταση απόψεων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ακολουθήσω λοιπόν τη σύσταση του συντονιστή του ΕΛΚ να ψηφίσουμε την πρόταση της κ. Κρέη. Θα κάνετε λοιπόν ψηφοφορία επί της διαδικασίας, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι λέει η Πρόεδρος, όπως είπα, θα ψηφίσουμε την πρόταση που υποβάλλει η κυρία Κρέλ. Να αλλάξει δηλαδή η σειρά των ε, τροπολογιών, πώς θα ψηφιστούν δηλαδή. Και θα το κάνουμε ηλεκτρονικά για να αποφευθεί οποιαδήποτε παρανόηση. Θα ψηφίσουμε δηλαδή εάν υποστηρίζουμε την πρόταση της κυρίας Κρέλ να ψηφιστεί πρώτη η τροπολογία, η συμβαστική τροπολογία των σοσιαλιστών. Εάν, εάν πείτε ναι, υποστηρίζετε την Κωνσταντσε Κρέλ. Αν όχι, τον εισηγητή. Ορίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. 26 υπέρ 19 κατά. Που σημαίνει ότι αλλάζουμε την σειρά της ε, ψηφοφορίας. Όπως το ερμηνεύω εγώ αυτό, σημαίνει ότι ψηφίζουμε πρώτα την συμβιβαστική 12 των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τις παραγράφους 21 και 23 που καλύπτει Καλά, ξέρετε τέλος πάντων τι ψηφίζουμε, το βλέπετε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ναι, ναι, αρχίζει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Πέρας. 27 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Τώρα λοιπόν Τώρα προχωρούμε λοιπόν στην 257. Α, εκπίπτει αυτή μου λέτε. Μια στιγμή πρέπει να ελέγξουμε. Συμβαστική 13. Συμβαστική 13. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ακολουθεί ...276... ...τροπολογία 276 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...277 και 78... ...εκπίπτουν έτσι δεν είναι... Συμβιβαστική τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 302, 302 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 313 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά παρακαλώ σηκώνετε καλά τα χέρια 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 και 19 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 3-20 υπέρ κατά αποχές 321 υπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3-22 μια στιγμή 3-22 υπέρ κατά απορρίπτεται 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 330 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 332 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 233 υπέρ κατά απορρίπτεται 334 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 16 Α, η κυρία Κρέλ ε, επ' αυτού μια διευκρινιστική ερώτηση δεν ξέρω πώς ακριβώς είχε διαμορφωθεί η συμβαστική τροπολογία. Στην τελευταία συνάντηση των, εισηγητών, ο των συντονιστών μάλλον, είπε ο εισηγητή ότι πρόκειται να αφαιρέσει την πρώτη φράση τη συμβαστική τροπολογία, διότι είναι αντίθετη με τι συνθήκε. Αυτό έχει συμβεί, έχει όντω αφαιρεθεί. Ο κύριο Πίπερ. Το πρώτο μέρος που αναφέρεται στα κριτήρια σταθερότητας έχει διαγραφεί. Το δεύτερο μέρος έχει μείνει, αν και είναι διατυπωμένο υπιότερα. Η κυρία Κρέλ. Μιλούμε για την συμβαστική τροπολογία 16 για το πρώτο μέρος που λέει για την συγχώνευση ταμείων που, ε, κονδυλίων που πηγαίνουν για ε, περιφερειακή πολιτική και συνοχή. Αυτό επρόκειτο να διαγραφεί, αλλά δεν ξέρω αν έχει διαγραφεί όντω. Βλέπω εδώ ότι δεν έχει τροποποιηθεί. Θα ρωτήσω, θα ρωτήσω τον σύμβουλό μου γιατί όχι, διότι έτσι είχε συμφωνηθεί ότι θα διαγραφεί το μέρος αυτό. Είστε διατεθειμένος να κάνετε προφορική τροπολογία τότε, επ' αυτού. Προτείνω, μου λέει και ο σύμβουλός μου, ότι αυτό που έχω μπροστά μου δεν είναι η τελευταία εκδοχή. Εγώ θα έλεγα η πρώτη φράση απλώς να φύγει, εκεί όπου αναφέρεται για διάλυση ή συγχώνευση. Το πρώτο λοιπόν αυτό μέρος να διαγραφεί, το δεύτερο να διατηρηθεί. Άρα η τροπολογία 16 λέει ότι τα ταμεία, αυτό, αυτή θα είναι η αρχή της ε, συμβαστικής τροπολογίας. Το θεωρούμε προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 16 όσο τροποποιήθη προφορικά. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική 16 όπω τροποποιήθη, ποιο είναι κατά. Αποχέ. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Έλεγχο. Θέλει κάποιο να ελέγξουμε τη συμβαστική 16. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη 16. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία μια ψήφος διαφορά 21-20 δίκιο είχατε που ζητήσατε τον έλεγχο αλλά εγκρίνεται Πάμε στην 3.47 προχωράμε. Έχουμε ακόμα πολλές. 3.47 υπέρ. 3.47 κατά. Αποχές εγκρίνεται. 349 καταπίπτει. 350, 350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 351 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 352 που τροποποιήθηκε είναι κάποιος κατά της τροποποίησεως όχι 352 τροποποιημένης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 353 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 355 υπέρ κα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 356 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 366. 366 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 367 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω, ας γίνει έλεγχος για την 367. Ξεκινά ο έλεγχος. 367. αρχή η ψηφοφορία. απορρίπτεται και μεγάλη διαφορά 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Η Ελίζαμπετ Στρέντερ έχει προφορική τροπολογία. Ναι. Έχω προφορική τροπολογία όπως συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις για τη συμβαστική 18 γραπτός διανεμήθη το κείμενο και προστίθεται εντός του συμβιβασμού τονίζεται η συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στις πρωτοβουλίες που, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι αποδοτικές ε, και να ληφθεί υπόψη και ο στόχος που υπάρχει για τους βιώσιμους, για τους βιώσιμους στόχους. Συμφωνείτε με την τροπολογία, είσαστε κατά. Ο εισηγητής είναι κατά. Αν είναι κατά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Ο εισηγητής είναι κατά λέτε. αυτό το θέμα, ο όρος flagship, οι εμβληματικές πρωτοβουλίες, ίσως είναι καλό να αναφερθούν. Απορρίπτει το ΕΛΚ την προφορική τροπολογία. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με αυτή την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 384 384 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 385 υπέρ κατά αποχές για την 385 πρέπει να ελέγξουμε δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα ξεκινάει η ψηφοφορία ο έλεγχος για την 385 τέλος απορρίπτεται 386 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται είσαστε κάπως σκόρπιοι και είναι δύσκολο να κρίνω νομίζω ότι εγκρίνεται θέλετε α εντάξει δεν χρειάζεται να λέξουμε. εγκρίνεται λοιπόν 387 κατά αποχές απορρίπτεται η 388 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 390 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω για την 390 είναι άγνωστο πρέπει να γίνει έλεγχος για την 390 ξεκινάει η ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται 391 υπέρ υπέρ 391 κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 405 πάμε τώρα 405 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 407 υπέρ κατά αποχές 407 ας γίνει ένας έλεγχος ξεκινάει τώρα όλες οι ομάδες είναι υπέρ άρα εγκρίνεται 407 εγκρίνεται 408 υπέρ κατά δεν είναι ξεκάθαρο έλεγχος για την 408. Απορρίπτεται. 409 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 410 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 412 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 413 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 415 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 416 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 418 υπέρ κατά θα γίνει έλεγχος για το 418 4-18 ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος απορρίπτεται 419 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 420 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 421 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος της 421 η 421 έλεγχος πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με διαφορά μίας ψήφου. 422 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 424 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 423 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα του 423. Θα κάνουμε ένα έλεγχο 423 πέρας Α, απορρίπτεται 425 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 426 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 427 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 428 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 429 υπέρ κατά έλεγχος για 429 ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 441 που τροποποιείται προφορικά είναι κάποιος που είναι εναντίον της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ποτέ δεν διαφωνείτε, οπότε σοκαρίστηκα. Λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε, 441. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 442. Υπέρ. Λάσλο. Λυπούμε, άκουσα τέσσερα από τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται είναι ότι η απασχόληση δεν έχει, δεν ξέρω αν καλύπτεται ή όχι. Μπορούμε να επανέλθουμε το θέμα το στην Ολομέλεια και δεν θα υποβάλω σχετικά προφορική τροπολογία. Τώρα θα επανέλθω στην ε, Ολομέλεια. Μένει ω έχει. Λέει η πρόεδρο, ναι, είναι η απάντηση. Ψηφίζουμε το 442 με τι πληροφορίε που μα έδωσε ο Λάσλο. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ είναι κατά. Θα ελέγξουμε την 442, γιατί δεν ξεκάθαρο. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται άρα είναι περίπου μοιρασμένες ψήφους λοιπόν συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μισό λεπτό να κάνουμε μια άκρη εδώ we vote the first part. So we go. No, but this the second on the first part. Okay, so we vote, now we go to... Πάμε στην 448 και ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα που έχει τροποποιηθεί με προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πάμε στη βαστική 22, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 461 461, Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 462, Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 465 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 464 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε τη 464 έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά τέλος Απορρίπτεται. 466 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι 468 και 69 είναι ταυτόσιμες τις ψηφίζουμε μαζί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πρέπει να γίνει έλεγχος για να είμαι σίγουροι Λοιπόν, ψηφίζουμε την 468 και 469 ηλεκτρονικά. Ξεκινά τώρα ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Εγκρίνονται. 470 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 472 υπέρ. 472 κατά. Αποχές εγκρίνεται μάλλον έλεγχος στα γρήγορα για 472 άρχεται η ψηφοφορία ο έλεγχος 472 Τέλος. Κάποιοι δεν ψηφίζουν. Δεν θέλουν, φαντάζομαι. Με τρεις ψήφους διαφορά. Εγκρίνεται. 473 υπέρ κατά δεν σηκώνετε το χέρι σας δεν σηκώνετε το χέρι σας το σηκώνετε ανάμεσα στο υπέρ κατά και δεν ξέρω είσαστε υπέρ κατά άρα πρέπει να γίνει έλεγχος για 473 ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 4,74 καταπίπτει και πάμε 4,75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,79 υπέρ κατά αποχές νομίζουμε ότι απορρίπτεται 280 Ε, Συνάδελφοι, έχουμε την 141 πρέπει να ψηφίσουμε μετά την 504. Ποιος είναι υπέρ, δεν ξέρω τι προβλέπει ο δικός κατάλογος, αλλά μετά την 504 στο, στο κατάλογο βλέπω την 141 τροπολογία. Αυτή πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. 141. Μπορούμε να ψηφίσουμε παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. 505. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 506 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 507 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 508 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 509 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 510 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 27 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 519 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται. 521 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 522 υπέρ κατά απόχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 522 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 523 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για την 524. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 525 ψηφοφορία κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 527. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Μόνο ο ή σήκωσε το χέρι του από το ΕΛΚ. Δεν είδα κανένα άλλο χέρι. Οπότε θεωρώ ότι το χέρι σας ανταποκρίνεται σε 17. Αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 527. Άρχεται η ψηφοφορία. «528» εγκρίθηκε προηγούμενη, κατά αποχές εγκρίνεται, «529» υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 530 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 531 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 532 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 533 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 533. ή μάλλον 534 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 535 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 536 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 537 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 538 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 557 557 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 558 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 559 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 560 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 560 την ψηφοφορία. Closed. Yeah, they don't vote, don't vote. Yeah, well, it's, it's rejected. Because ναι, ναι, Απορρίπτεται ναι. γιατί είναι ισοπαλία. Αλλά δεν ψήφισαν όλοι όσοι προβλέπονται. Ψηφίστε παρακαλώ όλοι για την 560. Χρειαζόμαστε 21 για να υπερψηφιστεί και ήταν 20. 560 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 44 έχουν γραφεί για ψηφοφορία, δεν ψηφίζουν όλοι. Τέλος. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται αυτή τη φορά με 23 ψήφους κατά. 521 και 63 επανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνονται. Αλλά στο το ελέγξουμε ηλεκτρονικά αν επιμένετε για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 561, 62 και 63. Τέλος και πάλι κάποιος δεν ψηφίζει, αλλά μάλλον κάποιος έφυγε, άφησε την κάρτα του. Now we go... ...569, ποιος είναι υπέρ, κατά, επαναλαμβάνω, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στα θεωρώντας. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Και θεωρώντας 1. Ψηφίζουμε μαζί ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά μάλλον εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6 άρχιτη ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 8 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται 3 και 10 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 και θεωρώντας 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 ε, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 ποιος είναι υπέρ κατά απο... ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 14 άρχεται ψηφοφορία Τέλος. Έγκρινεται. 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας τώρα, τροπολογία 16 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για την 28. Τέλος απορρίπτεται 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 37 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές Μάλλον απορρίπτεται. Δεν σηκώνουν τα χέρια τους. Πώς καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 41. η ψηφοφορία. The vote is... Τέλος. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Γρήγορα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 42, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ ε, κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για τι 48 άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται ή όχι. Μάλλον όχι, είναι ισοπαλία, χρειάζεται μία ψήφο παραπάνω. Απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, απόχέ, μάλλον απορρίπτεται και αυτή. Ή 50 τώρα, ποιο είναι υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 51, μάλλον 52, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ παρακαλώ τα χέρια ψηλά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στη δεύτερο, δεύτερο θεωρώντας από την Επιτροπή Απασχόλησης. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος του θεωρώντας 2. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θεωρώντας 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, πρώτο τμήμα από το 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 ή μάλλον 4 του 1 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το τέταρτο τμήμα του 1 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα του 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο ή μάλλον πρόταση 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται. 5, τροπολογία, πρόταση 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρόταση 6, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρόταση 12, άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα του 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μια στιγμή λίγο για να σκεφτούμε τα περαιτέρω. 21? Yes, 21. We vote. So we vote 21. Ψηφίζουμε την πρόταση 21, εκτός και αν κάποιος έχει διαφορετική γνώμη. Για το 21 υπάρχει πρόταση να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο πρώτα και αν απορριφθεί, για την παράγραφο 39 δηλαδή του αρχικού κειμένου, αν απορριφθεί τότε θα ψηφίσουμε την πρόταση 21. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, οπότε θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση 21. Ποιος είναι υπέρ. Who is against? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έχουμε μία μόνο τροπολογία που μπορεί να τρόπο. Δεν έχουμε μόνο μία τροπολογία για την 39 Έχουμε και την πρόταση 22. Αν εγκριθεί 22, τότε αυτή θα δικαταστεί στην παράγραφο 39. Η παράγραφος 39 έχει διαγραφεί όμως από το αρχικό κείμενο ψηφίζοντας κατά. Το καταλάβατε. Elizabeth Έχουμε τρεις δυνατότητες εδώ για το περιεχόμενο του Κοινωνικού Ταμείου. Η πρώτη είναι το αρχικό κείμενο της 39, η δεύτερη πιθανότητα είναι η σύσταση 21 και η τρίτη δυνατότητα η σύσταση 22. Το αρχικό κείμενο και 21 έχουν καταπέσει, έχουν απορριφθεί. Μας μένει το 22. Αν κάποιος θέλει να, να πει δύο λόγια για το περιεχόμενο του κοινωνικού ταμείου, θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της πρώτης 22. Εντάξει, είναι σαφές για το 39 και το 21. Θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε γιατί είναι ευαίσθητο το ζήτημα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρόταση 22, έρχεται ψηφοφορία. Closed. Τέλος. Απορρίπτεται και 22. we only vote, we only vote the first of these two of 24. Okay. The first part on. Okay. So now we move to the first part of. Πρώτο τμήμα του 24. So we go to the second. Δεύτερο για το 24. Το τελευταίο τμήμα καταπίπτει, ψηφίζουμε τα υπόλοιπα. Ποιος είναι υπέρ. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Την ξεχάσαμε πριν αυτή την πρόταση. other people from this delegation doing it. 25 we do vote, so we vote 25. Ψηφίζουμε την 25 τώρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε την 29. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, πρόταση 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πρόταση 4. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της πρώτης 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προτάσεις της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φύλων αιτιολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη D, δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, ε, υπέρ, κατά, αποχές, F, ε, σίγμα τάφ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, Z, G, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, ένα ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 2, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4 άρχεται η ψηφοφορία It's closed τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 6 υπέρ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 σήκωσα προς τα πάνω τα αντίχειρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και 15, 16, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 17, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά, 31 ψηφί υπέρ, 4 κατά, 9 αποχές. Συγχαρητήρια θερμά κύριε Πίπερ. Και πάμε στην έκθεση του Όλτριχ Βλασάκ. Mm. weaknesses as well. Έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Δεν είμαι τέλεια. So you didn't tell me. I'm sorry for... Δεν μου το είπατε. Λυπούμε που μου το είπατε μόνο τώρα. Πού είμαστε. 102 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε Αναθεωρώντας πρώτα στο 2 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται, η 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, αιτιολογική 4 υπέρ. Πρέπει να γίνει έλεγχος. Ελέγχουμε την αιτιολογική σκέψη 4. Υπέρ τη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 Στην τροπολογία 5 της ιδεολογικής σκέψης Α, η γραμματεία έπρεπε να αλλάξει τη σειρά. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι το πρώτο και το δεύτερο νομικά σαφές. Α, το νομικά σαφές, το legally clear. Το πρώτο τμήμα ξεκινά το εκτιμώντας, whereas. Έχει αλλάξει. Αυτό που ήταν πριν δεύτερο έχει γίνει πρώτο και το πρώτο δεύτερο. Ψηφίζουμε λοιπόν το, το, το, το πρώτο τμήμα που ξεκινάει με το εκτιμώντας, whereas. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται και πάμε στο νομικά ξεκάθαρο, legally clear, το δεύτερο τμήμα. Δηλαδή, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το ανθρωπολογία 7 υπέρ κατά αποχές Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 εδώ έχει ζητηθεί κατά τμήματα. Ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας κάνουμε μια επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της υπαριθμών 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Πω, πω, κοιτάξτε, απερίφθη. Με, με συγχωρείτε. Ωραία. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για το σύνολο της εκθέσεως αρχίζει η ψηφοφορία πέρας, πέρας, ναι, ναι, βεβαίως μια στιγμή, μια στιγμή Καλά, αν κάποιος καθυστέρησε θα προσθέσουμε την ψήφο του. Τώρα έληξε λοιπόν. Προχωρούμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διαταξής μας. what is the deadline? Yeah. Well, to be reminded of the time. No, wait a minute, wait a minute. Sorry, sorry, sorry. sorry. Except with my... Dear colleagues, yeah. Η πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, Γιάννη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα θυμάστε, ε, θα θυμάστε ότι δεν τελειώσαμε την συζήτηση της γνωμοδότησης του Γιάνν Όλμπριχτ για τον δημοσιονομικό κανονισμό, που είναι θέμα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να πω το εξής. Μα λέω κάπου κάπου σημαντικά θέματα και αυτό είναι από τα σημαντικά που σας λέω. Δεν τελειώσαμε λοιπόν την συζήτηση της ε, έκθεσης του Γιάνν Όλμπρεχτ για τον δημοσιονομικό κανονισμό που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της πολιτικής μας. Προτείνω λοιπόν αυτό που προτείνω μάλλον τώρα είναι να καθορίσουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 30 Μαΐου 12 το μεσημέρι και να δώσουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε διότι άλλη λύση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γιάνν, έχετε κάποια άλλη πρόταση, σύσταση. Μπορούμε ενδεχομένω να κάνουμε και μια έκτακτη συνεδρίαση με τον Γιάννη ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να προσέλθει, αν θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε αυτή τη συζήτηση. Όλμπριχτ. Τα ενδιαφερόμενα μέλη ας έλθουν σε επαφή μαζί μου πριν καταθέσουν τροπολογίε. Καλά, ας συμφωνήσουμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν τροπολογίε μέχρι την 20η Μαΐου και όσοι, κυρίω οι συντονιστέ επιθυμούν να συζητήσουν με τον Γιάν, α το πράξουν και αν κάποιο χρειάζεται έκτακτη συνεδρίαση με τον Γιάν, ο Γιάν είναι διαθέσιμο. Συμφωνούμε λοιπόν επ' αυτού. σα ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε εάν είναι κάποιο ακόμα από την Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή, ε, να έχει υπόψη ότι θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον Γιάννη, ο Γιάννη με αυτόν, γιατί τώρα έχουμε βέβαια και την ακρόαση που είναι πολύ σημαντική. Αρχίζει λοιπόν αμέσως η ακρόαση. Παρακαλώ πρώτα να καθίσετε όλες και όλοι. Ελπίζω οι εμπειρογνώμονες να είναι κοντά μας και τους απευθύνω το καλώς ορίσατε θα ακούσουμε πέντε, πέντε τοποθετήσεις για ένα σύστημα παροχής που βασίζεται στα αποτελέσματα και επιδόσεις στην πολιτική συνοχή. Θα σταματήσω αμέσως να μιλώ, αλλά παρακαλώ τους εμπειρογνώμονες να είναι το δυνατόν συντομότεροι να πούν αυτά που θέλουν, αλλά το δυνατόν συντομότερα, για να μας μείνει και λίγος χρόνος να συζητήσουμε. Χωρίς λοιπόν περισσότερα λόγια, ο ανεξάρτητος σύμβουλος κ. Μπέντ Πέριν της Διεθνούς Οργανώσεως Αξιολόγησης και Γενικός γραμματέα της Ευρωπαϊκής Εταιρεία Αξιολόγησης. Έχει το λόγο, αγαπητέ κύριε. with the papers, yes, it's But why they are trying to do it now? <laughs> I don't think he um, has... I think that uh, uh, Mr. Perrin didn't hear that I invited... Ίσως ο κύριος Περίν να μην άκουσε ότι του ε, δίνω τον λόγο. Ε, ας λάβει το λόγο ο κύριος Περίν και επίσης παρακάλεσα τους ε, και τις ομιλήτριες να είναι το δυνατόν συντομότεροι ώστε να προλάβουμε να κάνουμε και ερωτήσεις. Hello? Can, can you hear me? Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν συντομότερος. Θα αναφερθώ σε λίγα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης εκ των αποτελεσμάτων και τους σχετικούς δείκτες. Πρώτα, ορισμένοι περιορισμοί των δικτών η δυνατότητα κατάχρησής τους και οι δυνατότητες ελαχιστοποίησης αυτής της κατάχρησης. Θα γνωρίζετε βεβαίως ε, την ε, καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού με την έκρηξη της ε, δεξαμενής Deep Horizon. Η κύρια ευθύνη ήταν της εταιρείας εξορίξεως της Transocean στην τελική τους έκθεση είπαν ωστόσο ανεξάρτητα από τον τα, τραγική απώλεια ζώων το, στατιστικά το ιστορικό μας είναι καλό. Και έχουν λάβει και μεγάλα μπόνους για την ασφάλεια. Αυτό σίγουρα είναι ένας δείκτης που δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Οι δείκτες λοιπόν έχουν και ε, το αποτέλεσμα να διαστρεβλώνουν την απόδοση. Και βέβαια, αντί ε, να εξυπηρετεί τους πραγματικούς σκοπούς του το πρόγραμμα, προσπαθεί να ικανοποιήσει τους δείκτες σε ορισμένες, νομο, ορισμένες δικαιοδοσίες για να μειωθούν οι λίστες αναμονής στα νοσοκομεία ξεπετούσαν πρώτα τους ασθενείς που είχαν ε, μικροασθένειες και άφηναν τους άλλους. Άλλο φαινόμενο είναι το λεγόμενο της creaming. Για παράδειγμα για την παροχή υπηρεσιών σε ανάπηρους ανθρώπους οδηγεί στην πολύ έντονη ανάγκη που αισθάνεται το προσωπικό αυτό να παραγνωρίζει τις ανάγκες των πιο ε, βαριών ε, αναπηριών. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για τους δείκτες των συναλλαγών. Τι σημαίνει για παράδειγμα να χρησιμοποιείται ο δείκτης των, του αριθμού των απασχολούμενων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε καλές θέσεις απασχόλησης ε, με κάποια σταθερότητα ή και λιγότερο καλές δουλειές που ίσως καμιά φορά απασχολούνται μονάχα για πολύ λίγες ημέρες. Και το ίδιο για την αυταπασχόληση είναι άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες για παράδειγμα και εξαρτάται ποιους περιλαμβάνει κανείς το δείγμα και τι νόημα έχει ο δείκτης των εκπαιδευμένων προσώπων. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μια εκπαίδευση δύο ωρών χωρίς καμιά πραγματική αξία ή κάποιων άλλων οι οποίοι έχουν περάσει μια εκπαίδευση έξι μηνών που τους προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να καταλάβουν και θέσεις απασχόλησης που έχουν κάποια διάρκεια και στο μέλλον. Οι δείκτες βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ορθά αλλά ο δείκτης σας δείχνει απλώς μια ε, πρώτη εικόνα μπορούν περισσότερο να θέσουν ερωτήσεις οι δείκτες και δεν προσφέρουν εξηγήσει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να προσεγγίσουμε το θέμα με άλλα μέσα. Και το κυριότερο μήνυμά μου είναι ότι οι δείκτες έχουν μεγάλο δυναμικό κατάχρησης. Και κυρίως όταν υπάρχει άμεση διασύνδεση μεταξύ των οικονομικών και της επίτευξης των στόχων. Και επίσης προγράμματα προσφοράς επιβράβευσης που διασυνδέονται με προκαθορισμένους στόχους αντί να σκεφτεί ο κόσμος τον εντοπισμό των προβλημάτων και να δει τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Τώρα, τι σημαίνει αξιολόγηση εκ του αποτελέσματος η ένταξη των αποτελεσμάτων και ιδίω στην πολιτική συνοχή. Γνωρίζω τι σημαντικέ προσπάθειε που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αρμόδιε γενικέ διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι και γι' αυτό νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό με να το πετύχουμε σωστά. Πρώτα-πρώτα, η αξιολόγηση εκ των αποτελεσμάτων σημαίνει ότι ολόκληρα, ολόκληρο το σύστημα, όλα τα επίπεδα έχουν μια, ένα προσανατολισμό προς την επίτευξη αποτελεσμάτων διαχείριση βασισμένη στα αποτελέσματα και μέτρηση εκ των αποτελεσμάτων. Στην πραγματικότητα όμως όλοι ασχολούνται ε, με τον τρόπο μέτρηση των αποτελεσμάτων. Έχω εδώ και ένα έγγραφο που μπορώ να σας δώσω μετά. Αυτό που χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα είναι μια άποψη της accountability που να είναι πραγματικά για τον 21ο αιώνα και να εξυπηρετεί ε, τα δημόσια συστήματα. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στην ε, ανάληψη ευθύνης είναι κυρίως για να διαπιστώνεται πού κατευθύνονται οι εισρωές, χρήματα κλπ. Αλλά δεν εξυπηρετεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. που συνήθως είναι μέσα σε ένα περίπλοκο περιβάλλον πολιτικής. Εδώ χρειάζεται μια νέα ενατένιση της accountability και μια πορεία βασιζόμενη στα διδάγματα των εμπειριών. Και το ίδιο να είναι ε, υπεύθυνοι, να λαμβάνουν τις ευθύνες τους δηλαδή όσοι, ε, και, και να προωθούν την καινοτομία. Ένα σύστημα προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σημαίνει ότι μια δημόσια υπηρεσία καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα απρόβλεπτο ε, περιβάλλον πολιτικής και χρειάζεται να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν σε μια τέτοια στόχευση. Θα σας αφήσω το έγγραφο αυτό μετά, μετά από μια συζήτηση γενική ε, ε τράπεζα τράπεζας με την Παγκόσμια Τράπεζα και με άλλους εμπειρογνώμονες. Τονίζω ορισμένα από τα πιο σημαντικά πρόγευσαν από τη συζήτηση αυτή. Πρώτα, η αναγνώριση του γεγονότος ότι μια προσέγγιση εκ του αποτελέσματος είναι νέα προσέγγιση και πρέπει βέβαια να ανταποκρίνεται σε όλα τα, σε άλλα τα επίπεδα του συστήματος. Χρειάζεται σημαντική αλλαγή στον προσανατολισμό και αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται απτή δέσμευση από τα υψηλότερα επίπεδα της ε, διοίκησης και μετά σε όλα τα επίπεδα αλλά και εκ των κάτω διότι αν δεν υπάρχει αυτό δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή νοοτροπίας και καμία άλλη αλλαγή. Χρειάζεται Επίζει ότι αυτό δεν είναι εύκολο, χρειάζεται εκπαίδευση και υποστήριξη σε διάφορα επίπεδα και όχι μόνο στο κατώτατο επίπεδο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η προσέγγιση χρειάζεται να είναι στρατηγική, ώστε να έχει συγκεκριμένους στόχους και για την πολιτική συνοχή. Δεν υπάρχει τίποτε επαναστατικό σε αυτά που λέω, ούτε καν το έγγραφο αυτό έχει τίποτε επαναστατικό, βασίζεται στις βασικές αρχές της, της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Χρειάζεται επίσης να αναγνωριστεί πώς κινείται κανείς σύμφωνα με ένα σχέδιο, αλλά και γιατί. Χρειάζεται λοιπόν αξιολόγηση για να μπορείτε να γνωρίζετε πώς να κάνετε τα πράγματα καλύτερα. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και την ε, εκτίμηση του αν η, πορεία προς την επίτευξη των στόχων είναι ικανοποιητική. Εάν υπάρχουν άλλες επιπτώσεις εκτός των σχεδιαστησών και μια επικοδομητική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του μέλλοντος. Υπάρχουν Βέβαια, πολλές, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεων που αναφέρεται και σε αυτά που εξήγησα προηγουμένως και βέβαια που αυτά προσπαθεί να κάνει η πολιτική συνοχή. Συμπεραίνοντας, επενώ τις ε, προσπάθειες που γίνονται για μία εκ του αποτελέσματος αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής που χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και όχι απλώς εξυπηρέτηση κάποιων στόχων. Θα σταματήσω εδώ και θα περιμένω ερωτήσεις. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόκτωρ Κέρχαρτ από το Μίνστερ, από το, από το Σέντερφελτ. Λοιπόν, όσο πιο σύντομος μπορεί να είστε, μας δίνει το χρόνο να σας ρωτήσουμε Δεν Ευχαριστώ και για την εισαγωγή που κάνατε και για την προσκλησή σας. Το ερώτημα για την περαιτέρω εξέλιξη ενός συστήματος αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής έχει κέριο χαρακτήρα. Τίθεται τώρα ενώ υπάρχει το θέμα εδώ και μια εικοσαετία. Γιατί τονίζεται τώρα περισσότερο το θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μας απασχολήσει το ερώτημα αυτό. Βέβαια δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει αυτό. Το πρώτο ερώτημα είναι το σύστημα αυτό τι θα πρέπει να δείξει και σε ποιο επίπεδο. Αυτό που θα πρέπει να δείξει είναι ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές επιτυγχάνουν τους στόχους τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Και αυτό ε, τόσο σημαντικότερο γίνεται όσο πρόκειται για τη συνέχιση της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο όπου όλες οι χώρες μέλη αντιμετωπίζουν σημαντική δημοσιονομική πίεση, αναγκάζονται να περικόψουν δικά τους εθνικά προγράμματα, να ε, απαιτούν ε, περισσότερα εισπρακτικά έσοδα φορολογικά δηλαδή από τους κατοίκους των κρατιών τους Επομένως χρειάζεται και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία ε, εκ των αποτελεσμάτων αξιολόγηση των προσπαθειών. Γιατί μιλούμε σήμερα για το ζήτημα αυτό, για την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Διότι τα άμεσα, ε, οι άμεσε ενδείξει που έχουμε από επιστημονικές έρευνες είναι πολύ αδύναμες. Όχι βέβαια για το ότι, για το ότι πράγματι εκπαιδεύτηκαν κάποια πρόσωπα, πράγματι κατασκευάστηκαν κάποιοι αυτοκινητόδρομοι, αλλά η απόδοση της προσπάθειας κατά κεφαλή. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που δείχνουν είτε ένα αδύναμο θετικό μεν αποτέλεσμα ή καμιά φορά και μηδενικό. Άρα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που δείχνει δηλαδή ότι τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής είναι δύσκολο να μεταφερθούν σε ε, οικονομικά μεγέθη, να ε, ερμηνευτούν ως οικονομικά μεγέθη. Υπάρχει και ένας αριθμός παραγόντων που κάνουν το σύστημα πιο περίπλοκο και που ενδεχομένως παρεμποδίζουν ε, να μπορέσουμε να καταμετρήσουμε τις θετικές επιπτώσεις το ίδιο το σύστημα είναι περίπλοκο, έχουν αλλάξει σημαντικές παράμετροι, υπάρχουν και πολλοί τομείς των παρεμβάσεων, όπου γίνονται παρεμβάσεις δηλαδή, και όπου συχνά είναι δύσκολο να γίνουν κοινέ μετρήσεις. Το δεύτερο αναφέρεται σε αυτό που γνωρίζουν οι οικονομολόγοι, ότι υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες σχετικά με τη γνώση μας, τι δηλαδή συναπαρτίζει την περιφερική ανάπτυξη. Η θεωρητική συζήτηση εξελίσσεται γοργά, αλλά έχουμε λίγα στέρεα εμπειρικά δεδομένα στη βάση των οποίων να μπορέσουμε να πούμε να αυτές είναι εξελίξεις και αυτοί είναι οι παράγοντες που τις καθορίζουν. Και ένας ακόμα παράγοντας της περιπλοκότητας είναι η, η αντίθετη περίπτωση, υποθετικά δηλαδή, θα γινόταν αν δεν υπήρχαν τα διαθωτικά ταμεία κάτι που πρόκειται για μια στάνταρ τεχνική, αλλά αυτή η κατάσταση, δηλαδή της εκ του αντιθέτου, πρέπει πρώτα να οριστεί. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, θα ήταν μια ε, κατάσταση όπου οι χώρες μέλη δεν θα διέθεταν ε, ε, απολύτως κανένα κονδύλιο. Άρα και εδώ είναι προβληματική η προσπάθεια ορισμού του, της εκ του αντιθέτου αποδείξεως. Ε, ε, έχουμε λοιπόν και, το πρόσθετη, την πρόσθετη δυσκολία ότι είναι πολύ σύντομες οι προθεσμίες για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Μου ζητήσατε να πω λίγα και για την μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Διακρίνω ανάμεσα στα επίπεδα όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα, τα μακρομοντέλα, θα πρέπει να εφαρμόζονται στο συνολικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τα μοντέλα που ε, ε, χρησιμοποιεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μοντέλα Quest και τα μοντέλα που έχω αναπτύξει εγώ με συναδέλφους μου, το Hermin. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα τα οποία προέρχονται από την θεωρία της ανάπτυξης και μπορούν να είναι μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται είτε από τις χώρες μέλη είτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό της. Όλα βέβαια έχουν και πλονεκτήματα και μειονεκτήματα που δεν θα με απασχολήσουν εδώ. Όμως εάν τώρα μιλείτε για συγκεκριμένα προγράμματα ή για συγκεκριμένα μέτρα, τότε χρειάζονται άλλες μέθοδοι. Υπάρχει και ένας ολόκληρος αριθμός διαφορετικών ε, ε, μετρήσεων. Ξεκινάει με τις ομάδες ελέγχου, control matching. Αυτά έχουν πάρα πολύ υψηλές απαιτήσει και για τους συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται με τις μετρήσεις αυτές, με συνεντεύξεις με τα αρμόδια πρόσωπα στις διάφορες εθνικές διοικήσεις, με τους ε, δικαιούχους απολύπτες και ούτω καθεξής. Αλλά το monitoring, interview και matching δεν λένε τίποτα για την αποτελεσματικότητα ή αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής. Λένε κάτι μονάχα για το συγκεκριμένο μεμονωμένο μέτρο, το οποίο ενδεχομένως συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλετε να μάθετε κάτι για τις ευρωπαϊκές διαθωτικές πολιτικές συνολικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα μεθοδολογιών που να περιλαμβάνει και μάκρο μοντέλα και μικρο μοντέλα και το monitoring. Άρα δεν αρκεί χρήση μιας μονάχα μεθοδολογίας για να, μετρήσει, για να μετρηθεί μάλλον η αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Διαθωτικών Ταμείων. Και έρχομαι τώρα στον, στην, κύκλο πολιτικής που έχει έξι βήματα και όπου υπάρχει ένα σύστημα για τις ε, παρεμβάσεις και έτσι καθορίζονται και οι στόχοι εφαρμόζονται στο ε, σημείο 4 μετά η αποτελεσματικότητα και συνεκτικότητα των παρεμβάσεων και από αυτές ε, συμπεραίνεται περί των αποτελεσμάτων. Στο 5 μιλούμε για ένα σύστημα βασισμένο στις επιπτώσεις αλλά δεν μπορεί να βασίζεται παρά μόνο στα σημεία 2, 3 και 4 όπου καθορίζετε εσείς με ποιο τρόπο που θα παρέμβετε και πού ακριβώς. Άρα δηλαδή καθορίζετε τους στόχους και από τους στόχους προκύπτουν οι δείκτες και οι μέθοδοι αναλύσεως. Άρα σε αυτό το, το σύστημα ενός προσανατολισμού βασισμένου στα αποτελέσματα προκύπτει ο εντοπισμός των προβλημάτων και των κατάλληλων μέτρων και αυτά λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να καθοριστεί το σύστημα στην βάση της λογικής της παρεμβάσεως. Ο ορισμός των επιμέρους ε, στόχων είναι δύσκολος και είναι δύσκολος να μετρηθεί. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για να μην καταναλώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ισχύει το εξής. Μέχρι τώρα δεν έχουμε σχεδόν καθόλου συγκρίσιμα δεδομένα για τις διάφορες χώρες μέλη. Όλοι δε οι παράγοντες τους οποίους καθορίζουμε ως μεταβλητές των στόχων καθορίζονται από εξωτερικούς παράγοντες και είναι και εξειδικευμένοι αναχώρα και ποικίλουν αναχώρα. Εάν εξετάσουμε ένα σύστημα το οποίο περιλαμβανόταν πρόσφατα σε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που εξηγεί τον κύκλο αυτό πολιτικής, από αριστερά προς τα δεξιά θα δείτε ε, πάνω και αριστερά τις ανάγκες, μετά τις προτεραιότητες εφαρμογής, μετά θα δείτε την εικόνα των actual outcomes, των πραγματικών δηλαδή επιπτώσεων αποτελεσμάτων. Και δεξιά θα δείτε ένα μικρό κουτάκι στο οποίο αναγράφεται άλλοι παράγοντες other factors. Αυτοί οι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι βέβαια επηρεάζουν την εξέλιξη των παραμέτρων, των στόχων, είναι στην ουσία κυρίαρχα δεδομένα. Αυτά μπορείτε να τα εξετάσετε ως την ενατένιση κάποιου που βρίσκεται μέσα στην πολιτική συνοχή, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι περισσότερο έτσι, δηλαδή το μέγεθος των άλλων παραγόντων είναι κυρίαρχο Θα πρέπει να δείτε δηλαδή την εξέλιξη των επιδοτούμενων χωρών και περιφερειών. Εκεί οι άλλοι παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες, οικονομικές εξελίξεις καταστρέφουν στην πραγματικότητα πράγματα τα οποία έχουν χτιστεί σιγά σιγά μέσα σε δεκαετίες από τα διαθωτικά ταμεία. Και αυτά οφείλουν να ληφθούν υπόψη όταν μιλεί κανείς για την αξιολόγηση των διαρθωτικών ταμείων. Ποιες είναι τώρα οι επιπτώσεις και τα συμπεράσματα. Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να έχει κανείς πάντοτε υπόψη ότι χρειάζεται διάκριση των δύο αυτών α, ε, σημείων. Η επιρροή δηλαδή που ασκούν τα διαφορετικα και άλλα ταμεία από τους άλλους παράγοντες. Άρα η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να παρενοχληθεί ή και να καταστραφεί από άλλους παράγοντες και να καταλήξετε έτσι σε, διαφορε... σε... σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Απλές συγκρίσεις σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα πραγματικά αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γίνουν. Δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Δεν μπορείτε να συγκρίνετε δύο πράγματα μέσα στην εξέλιξη του χρόνου χωρίς να κάνετε ταυτόχρονα έλεγχο όλων των υπολείπων παραγόντων. Και κάτι ακόμη σημαντικό. Βραχυπρόθεσμα πολλά από τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων των διαθωτικών ταμείων δεν θα είναι ορατά. Πρωτίστως πρόκειται για την εφαρμογή και όχι για τα αποτελέσματα. Θα δείτε έργα από ένα συγκεκριμένο ε, την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι μακροπροθεσμότερα. Για παράδειγμα, ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ούτω καθεξής. Και υπάρχει επομένως σημαντική παρέλευση χρόνου μέχρι ότου υπάρξουν, γιατί στο περιφερειακό επίπεδο συχνά είναι 2-3 χρόνια η, ε, η περίοδος αυτή. Είναι λοιπόν πολύ φιλόδοξο να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα. Παρ' όλα αυτά εγώ το θεωρώ απολύτως απαραίτητο να, συνεχίσει, να συνεχιστεί η προσπάθεια, ωστόσο τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που κινούμαστε τώρα πλέον προς την ε, κατεύθυνση ενός συστήματος τέτοιου αξιολόγηση εκ του αποτελέσματος που δεν σημαίνει και κανένα ριζοσπαστικό νεωτερισμό αλλά μια περαιτέρω εξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος το οποίο πάντοτε λειτουργήσε στη βάση προκαθορισμένων στόχων, είναι ευκολότερο, όπως είπα και πριν, να εξετάσει κανείς τα προβλήματα για να αντιληφθεί ποια είναι η λογική της παρέμβασης και τι νόημα έχει να γίνονται λάθος παρεμβατικά μέτρα τα οποία δηλαδή εξυπηρετούν λάθος καθορισμένους στόχους και έτσι πετάμε τα χρήματα από το παράθυρο. Γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των μεταβλητών των στόχων. Και από αυτό προκύπτει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρότερη και ιδίω στο μικρό επίπεδο και η προσέγγιση της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο είναι σίγουρα η ορθή, ο σωστός δρόμος. Στο μάκρο επίπεδο γίνεται αυτό ούτως ή άλλως. Δεν γίνεται και διαφορετικά και στην ουσία χρειάζεστε και τις δύο μεθόδους για να μπορέσετε να πείτε κάτι τι σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των, ευρωπαϊκών, των παρεμβάσεων μάλλον των Ευρωπαϊκών Διαστατικών Ταμείων. Το γεγονό ότι υπάρχει αυτή, αυτό το χρονικό κενό ανάμεσα στις ε, παρεμβάσεις και στη δημοσίευση είναι διότι δίνεται περισσότερη, αποδίδεται περισσότερη αξία στην ε, διάρθρωση των παρεμβάσεων και λιγότερο στην αποτελεσματικότητά τους. Διότι τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να έχουν μακροπροθεσμότερη ε, ενέργεια. Και αυτή μπορεί να μετρηθεί μόνον εφόσον επιτρέψετε να παρέλθει χρόνος ώστε να αρχίσουν να ενεργούν τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Ας μιλήσει ο πρώτος που έχει συνοπεκλωτική εμπειρία, η κυρία Έλενα Ταλιάνη, χάρη, εκπροσωπεί τις περιφερειακές αρχές της Εμίλια Ρωμάνια, οπότε σας παρακαλώ να παρουσιάσετε τις ε, απόψεις σας. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα βασιστώ σε αυτά που είπε ο καθηγητής που αναφέρθηκε σε πάρα πολύ σωστό θέμα που αναφέρθηκε στην περίπλοκη φύση της πολιτικής συνοχής και χρησιμοποιώ εγώ μια προσέγγιση που δεν είναι θεωρητική του καθηγητή γιατί εγώ είμαι νομικός ε, όμως για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σημαντικό αυτό το στοιχείο, διότι περίπλοκο χαρακτήρα τη πολιτική συνοχή συμπίπτει με το χαρακτήρα τη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Που γνωρίζουμε ότι ενώ άλλε πολιτικέ ε, έχουν ένα στόχο προκαθορισμένο, συγκεκριμένο, που περιγράφεται, πλαισιώνεται, εδώ έχουμε σχετικιστική ε, προσέγγιση και πρέπει να υπάρχει δυναμική ισορροπία μεταξύ περιφερειακών αναπτύξεων και θα πρέπει να μειωθεί αυτό το κενό τη διαφορά που υπάρχει σε εδαφικό επίπεδο. Πέραν αυτού, περιφερειακό εγενή χαρακτήρα αυξήθηκε με την εισαγωγή της συγκεκριμένης συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως του περασμένου έτους της έννοιας της εδαφικής συνοχής που πρέπει να την έχουμε υπόψη διότι καθιστά δεσμευτική πολύ ισχυρή την απέτηση να δοθεί μια πραγματική εδαφική διάσταση στην πολιτική που ε, εφαρμόζεται στις περιφέρειες. Αυτό το τον περίπλοκο χαρακτήρα προσφέρεται και ιστορική καιρή που περνάμε τώρα που όλοι συζητούμε και σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά όλα τα βήματα που γίνεται συζήτηση για την περίοδο που περνάμε. Δεν θα σταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά την ε, επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωρίζουμε ότι βασίζεται στα, στα achievements, στα επιτέγματα. και ε, εστιάζεται επίσης επί της ε, ποιότητας του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου που είναι κλειδί για πραγματική αποτελεσματικότητα ε, της πολιτικής της συνοχής και όλα αυτά βασίζονται στο ότι, δε, ότι γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα αξιολογήσεως της παρούσας πολιτικής συνοχής ε, δεν ήταν ικανοποιητικά είναι ποσοτικά, δεν είναι ποιοτικά, είναι μερικά, δεν είναι συγκρίσιμα, όλα αυτά τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, η, η, πρόταση βασίζεται, βασίζεται πρόταση επιθεωρητικής βάσεως. Εκεί βασίζεται το πακέτο της, είναι μια πρόταση που ξεκινώντας από αυτή την έννοια που προανέφερα προτείνει μια προσέγγιση για την ανάπτυξη που ε, ακολουθεί την εδαφική διάσταση για να μειωθούν οι ανεπάρκειες και να, να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μένει η πολιτική συνοχής ε, θεωρείται σαν ιδεώδης βάση για να γίνει ποιοτικό άλμα στον αφορά τον προγραμματισμό. Αυτό όμως χρειάζεται κάποιες αλλαγές σημαντικές. Και ήδη γίνει και μια μικρή αξιολόγηση ε, όπως έκανα εγώ ε, των δεχόμενων συνεπειών που θα μπορούσε να έχει αλλαγή της προσέγγισης καθορίζοντα της πολιτικής ε, που ακολουθούνται ε, πόσο θα είναι παραγωγικές ε, ποιοτικά και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αν λοιπόν η αξιολόγηση ε, ε, που δεν, είναι, δεν γίνεται πολύ συχνά και εμποδίζει σωστέ επιλογές ε, μειώνει την αποτελεσματικότητα και αυτό είναι προβληματικό και μειώνει την αποδοτικότητα της πολιτικής συνοχής. Δεν θα σταθώ τώρα στα, στο τι είναι το νέο σύστημα που προτείνεται διότι ήδη οι πρώτοι δύο συνάδελφοι, οι δύο αγορητές μάλλον τα ανέφερα καλύτερα θα έλεγα ότι όλα βασίζονται σε ένα ίδιο πλαισίωσης λογικής που πρέπει να είναι ε, και χρονολογικά συντονισμένες για την πολιτική απόφαση και την επιλογή των μέσων για την διαχείριση της πολιτικής. Σημαίνει αυτό να μπορεί να αλλάξει η πολιτική, να μπορεί να προσαρμοστεί, να συγκριθεί και να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση από εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις σε κάποια στάδια και θα πρέπει ε, να ε, υπάρχει και ένας έλεγχος και να, να κρίνουν οι διευθύνοντες αυτή την ε, όλη προσέγγιση. Υπάρχει πολλαπλή διάσταση που αυτό είναι κάτι επί το οποίο συμφωνούμε κατά πολύ. Λοιπόν, βλέποντα την περιφερειακή προσέγγιση στο θέμα, από αυτήν η δική μα εμπειρία, βλέπουμε σε μια τέτοια αλλαγή όπως διερευνάται μεγάλη δυνατότητα να καταλήξουμε σε συγκεκριμένη ε, ανάληψη ευθυνών του δημόσιου φορεί σε ό,τι επίπεδα τη ε, κυβερνήσεω, ξεκινώντα από το δικό μα επίπεδο το περιφερειακό και σε όλε τι φάσει τη πολιτική, την απόφαση, την εφαρμογή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και στο τέλο και το feedback και το νέο κύκλο που αυτό καθορίζεται σαν όνεση η ιδιοκτησία της πολιτικής από πλευράς εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις από το δημόσιο τομέα και προς τα έξω σαν ε, ε, λογοδοσία, accountability, δηλαδή να μπορεί και το κοινό να βλέπει πώς κινούνται αυτοί οι φορείς. Υπάρχουν στενοί θεσμοί μεταξύ της απόψης πολιτικής και των μέσων που χρησιμοποιούνται για να γίνεται η διαχείριση της πολιτικής. Χρειάζεται ένα έλεγχος, χρειάζονται δύο συστήματα λοιπόν ποιοτικά ε, ε, και τα άλλα που προσθέτουμε εμείς είναι ανανεωμένη προσοχή στην κλίμακα την δαφική στην κλίμακα εκείνη στην οποία λαμβάνονται αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο. Κατά την άποψή μα είναι αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου που στην πραγματικότητα πέρα από το περιεχόμενο τεχνικό αυτά αφορούν αποκλειστικά πολιτικές πτυχές, διότι αφορούν την χρήση μιας, την εφαρμογή μιας πολιτικής επιλογής. Τόσο αφορά τις αλλαγές που αναμένονται, εμείς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα νέο στατηγικό πλαίσιο που τίθεται για να δοθεί μεγαλύτερη ισχύ στη στατηγική επιλογή εκ των άνω, η αρχή της συγκέντρωσης, η τάση της ολοκλήρωσης των διαθετικών ταμείων και μετά δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συμβάσεις ε, σύμπραξης για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις που προφανώς σύμφωνα ανάλογα με την περιφέρεια πρέπει να εξετάζονται να... πώς οι κεντρικοί φορείς ε, είναι σημαντική. Αν εκεί στα μέρη αυτά που στη διέλευση από τις επιλογές στρατηγικές και τα λειτουργικά προγράμματα ε, αυτοί οι κόμβη θα πρέπει να, είναι, να, να εφαρμόζονται επιθελοντικής βάσεως. Ε, λοιπόν, ξοδεύονται το χρήματα την πολιτική συνοχή. Το ξέρετε εσείς καλύτερα από εμά. Ξέρετε τα στοιχεία. Και εσείς θέλετε να ξέρετε πώ θα χειριστήκαμε με τα χρήματα σε περιφερειακό επίπεδο. Και χρειάζεται αυτή η σωστή διασύνδεση. Ευαίσθητο θέμα είναι το εξή. Πρέπει να είναι ένας τόπος εκεί, πρέπει να υπάρχει τόπο όπου καθορίζονται συγκεκριμένα λεπτομερώ τα μέσα που πρέπει να χειρίζονται τι πολιτικέ και τι παρεμβάσει τι συγκεκριμένε. και πιστεύω ότι μέσα στη συμβάσει σύμπραξης θα πρέπει να αναλαμβάνεται μια υποχρέωση και πλευρά των μελών και μόνο, αλλά πλευρά των περιφερειών να ετησίω ανάλογα με την ανάπτυξη πολιτική συνοχή να υπάρχει μια σχετικοποίηση στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμιση ενόψη τη Ευρώπη του 2020. Διότι είναι εκτό στρατηγική Ευρώπη του 2020 οι περιφέρειε. Αλλά ζη... πώ θα ευθυγραμμιστούμε διαφορετικά όμω. Ένα τρόπο είναι αυτό. Να είναι ξανά ενεργέ οι περιφέρειε στη διαμόρφωση στρατηγική Ευρώπη του 2020, αλλά να υπάρχει ε, μεγαλύτερη πολιτική ευθυγράμμιση στην πολιτική συνοχή συναρτήση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην Ευρώπη του 2020. Χρειάζεται έλεγχο, αξιολόγηση, τα είπαμε αυτά Υπάρχει αρχή τη απλούστευτη που είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών και βέβαια πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη προσοχή να αποφευχθεί να γίνει επανεθνικοποίηση που σε χώρε όπω είναι η δική μου Ιταλία θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα, τεράστια προβλήματα, κυρίω όσον αφορά στην πολιτική τη συνοχή που έχει μια ιδιαίτερη φύση, όπω αυτή που προανέφερα. Λοιπόν, αυτή η αλλαγή όπω τη βλέπουμε εμεί είναι όχι μόνο τεχνικώ εφικτή, ε, διότι σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε όλα τα επίπεδα των θεσμών που χειρίζονται ήδη αυτή τη στιγμή την πολιτική συνοχή, υπάρχει η δυνατότητα η διοικητική, υπάρχει επίση και επίγνωση αυτή τη αλλαγή. Δεν είναι μόνο σκόπιμο και χρήσιμο, διότι τώρα είναι στιγμή να μιλάμε για μια αλλαγή που αφορά τον επόμενο κύκλο χωρί να κάνουμε τι αλλαγέ εν μέσω εδώ, αλλά για μα είναι όχι μόνο συζητάμε, ε, είναι ανα... πρέπει να γίνει, αλλά είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο. Η πολιτική συνοχή είναι υπέρ των περιφερειών. Είναι γίνεται για να γίνει σωστή εκμετάλλευση των ιδιαιτεροτήτων. Αν δεν υπάρχουν προσμετρήσιμε συγκεκριμένες συνέπειες, συγκρίσιμε για να είναι αναποτελεσματική, άχρηστη πολιτική. Αν οι περιφέρειες δεν μπορούν να δουν τα ωφέλη, ε, δεν έχει νόημα να ασκεί κανεί ε, πολιτική συνοχής. Υπάρχει κι άλλο κίνδυνο ε, βέβαια των εσφαλμένων αλλαγών ή να μην γίνει καμία αλλαγή. Έναντι αυτών θα έλεγα ότι ο κίνδυνος αυτός ε, δεν θα πρέπει να εμφισταθεί. Είναι κάτι που μπορούμε να αποδεχθούμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα, τα θεσμικά, ε, αλλά βλέπουμε βασικά ότι τι πρέπει να γίνει από πλευρά εξορθολογισμού, αναδιοργάνωση και επιμερισμού των διαφόρων μοντέλων. Να χρησιμοποιηθούν δομέ που ήδη υπάρχουν και που ήδη εργάζονται όσον αφορά την πολιτική τη συνοχή. Εμεί πιστεύουμε λοιπόν ότι η διοικητική δυναμικότητα όσον αφορά τι δομέ ήδη υπάρχει δεν θέλουμε να προσθέσουμε πόρους, δεν χρειάζεται αυτό ή να συνοδευτεί η δομή ή να πάνε παράπλευρα δομές. Χρειάζεται να επανεξεταστούν, να δούμε ποια προσέγγιση χρειάζεται, ποιο μοντέλο χρειάζεται που εξυπηρετεί όλους για να δουλεύουν καλύτερα με διαφορετικό τρόπο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ένας άλλος τρόπος, άλλο πράγμα που βλέπω εγώ, σχέση είναι το commitment. Χρειάζεται λοιπόν αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει πολιτικέ να γνωρίζουν την εμβέλεια που συνεπάγεται η αλλαγή προσέγγισης ε, στο πολιτικό επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα, θα ανταποκρίνεται σε αποφασιστική αλλαγή όσον αφορά την ποιότητα και την αποδοτικότητα της πολιτικής της ε, συνοχής. Και λοιπόν κλείνω λέγοντας ότι αν θέλουμε μια αποτελεσματική πολιτική, ένα σύστημα που είναι που οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και δίνει καλύτερες επιδόσεις, είναι πιο ποιοτικό, ε, μπορεί να είναι ποσοστική σημασία αν γίνει σωστά σε επίπεδο περιφερειακό, εδαφικό και να λάβουμε υπόψη ότι οι εδαφικέ συνέπειε θα πρέπει να είναι ποιοτικέ, ποσοτικέ και θα πρέπει να μπορούν να είναι συγκρίσιμα αποτελέσματα και να μπορεί να γίνει αποτίμησή του. Ε, νομίζω ότι τα είπα όλα. Εδώ είμαστε υπέρ αυτή τη αλλαγή προσέγγιση. θέλουμε ότι είναι ριζοσπαστική και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε. Ε, νομίζω ότι τα είπα όλα. very uh, Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Υφυπουργό της ε, Λετωνίας, τον κύριο Αλεξάνδρης Αντόνοφς από τη Ρίγα, για να μας παρουσιάσει τις δικές του απόψεις. Ε, και εγώ όντως κατάγομαι από τη Ρίγα, αλλά κανονικά δεν πρέπει να το λέω, ε, λέω από τη Λετωνία. Ε, ζητήθηκε η εθνική σκοπιά για το σύστημα που προσανατολίζεται περισσότερο στι επιδόσει. Ξεκινάω από ένα θεωρητικό θέμα. Σε περίπτωση περιορισμένων ικανοτήτων, γιατί πάντα τέτοιε έχουμε, περιορισμένα διοικητικέ ικανότητε. υπάρχει αυτή η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ των ελέγχων και της ανάλυσης ε, των αποτελεσμάτων μιας πολιτικής θα πρέπει να δούμε πού μας οδήγησε αυτή η πολιτική και αυτή η επιλογή μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια. Στις τρεις τελευταίες περιόδους προγραμματισμού, γιατί είναι αυτή η μόνη ιστορική αναφορά που έχουμε εμείς στη Λετωνία, είδαμε ότι το σύστημα αυτό του, της πολιτικής συνοχής επικεντρώθηκε περισσότερο στους ελέγχους εκ των προτέρων και όχι στα αποτελέσματα στους ελέγχους με βάση τις πληροφορίες, το input. Και μάλιστα οι προτινόμενες τροπολογίες στο δημοσιονομικό κανονισμό θα είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή τη λάθος κατά τη γνώμη μου την εσφαλμένη κατεύθυνση. Είναι ένα επιπλέον βήμα προς τους ελέγχους ε, της ε, του input των στοιχείων που δίνονται εκ των προτέρων παρά ένα βήμα προς την κατεύθυνση το, της αξιολόγησης εκ των αποτελεσμάτων. Με βάση δηλαδή τις επιδόσεις. Θα πρέπει η επιλεξιμότητα να περάσει από τους ελέγχους του input προς την υλοποίηση των αποτελεσμάτων. Από μαθηματική άποψη δηλαδή τα κονδύλια που λαμβάνουν οι περιφέρειες ή τα κράτη-μέλη να είναι ε, με τα αποτελέσματα που υλοποιούν σε αντίθεση με την ισχύουσα κατάσταση που τα κονδύλια που λαμβάνουν τώρα είναι ε, αντίστοιχα με την ικανότητα των λογιστών ε, των αρμοδίων να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να ξοδέψουν το α ή το β ποσό. Και ας ε, προσπαθήσω να τεκμηριώσω με επιχειρήματα αυτή τη θέση. Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα και να εφαρμοστεί προϋποθέτει μεγαλύτερη καλύτερο και ενισχυμένο ρόλο της αξιολόγησης και, της, ε, και μια αναλυτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιούν τα κράτη-μέλη. Σε περίπτωση όμως περιορισμένης οικονομικής ε, δυνατότητας, όπως, ισχύει, συμβαίνει, θα πρέπει να, μειωθεί η, το βάρος των ελέγχων και της αναφοράς, κάτι που έχει μεγάλη βαρύτητα στο ισχύο σύστημα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι οριζέντες ε, πολιτικές και το σύστημα δημόσιων προμηθειών ε, αφαιρεί από τη διοίκηση της το χρόνο και το προσωπικό που θα μπορούσαν να αφιερώσουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τις οριζόντιες πολιτικές. Μιλούμε για μια πολύ διαφορετική δηλαδή προσέγγιση από αυτή της πολιτικής συνοχής. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση των Βρυξελών, πολλές γενικές διευθύνσεις έχουν επιλέξει να αφιερωθούν στην ενίσχυση των Γενικών Διευθύνσεων για τα Διευθυντικά Ταμεία. Γενική Διεύθυνση ε, Άγκρη, Ρίτζιο, ε, Θαλασσών ενισχύουν τις πολιτικές τους που εμπίπτουν στις ε, εντολές άλλων γενικών διευθύνσεων. Αυτό βέβαια βολεύει πολλές ε, διευθύνσεις και είναι προς όφελός τους, αλλά δημιουργεί πρόβλημα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν θέλω να φανώ μηδενιστής, ούτε είμαι πολύ απεσιόδοξος για τις οριζόντιες πολιτικές και την ενιαία αγορά. Αλλά είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να επιβαρύνουμε την πολιτική συνοχής με την, με την εφαρμογή και των άλλων οριζόντιων πολιτικών που κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζονται αλλού. Αν μια γενική διεύθυνση πιστεύει, πιστεύει ότι δεν εφαρμόζονται οι έλεγχοι των κρατικών ενισχύσεων, θα πρέπει να διορθώσουν την κατάσταση στα πλαίσια της δικής τους εντολής και όχι να την παραπέμπουν στην πολιτική συνοχή. Αν θεωρούν ότι ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει σωστά τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, τότε θα πρέπει να το εξετάσουν ε, στα πλαίσια της συγκεκριμένη πολιτικής και όχι να τα επιρρύπτουν όλα στην πολιτική συνοχής. Προχωρώντας τώρα περαιτέρω στο θέμα του προγραμματισμού και στη φάση της στρατηγικής, πιστεύουμε ότι ακράδαντα ότι και τα κρατημέλη και οι περιφέρειές τους πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να επιλέγουν τις προτεραιότητες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και μετά να συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φυσικά να συμφωνούν και για τα αποτελέσματα που θα επιδιώξουν και θα... αποτελέσματα που θα αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω χρηματοδότηση του προγράμματος σε μεταγενέστερες φάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τους στόχους που θα πρέπει να έχουν τα προγράμματα, θα πρέπει να είναι φυσικά ευφύς, ε, μάλλον SMART, Specific Measurable Attainable Relevant και Time Bound, ε, Αυτό είναι τα, το ακρονίμιο. Θα δούμε τι γίνεται μετά με το input. Επίσης θα πρέπει να επικεντρώνουμε τους δείκτες ε, πολύ λιγότερους αλλά πιο συγκεκριμένους και εδώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μοιράσει ένα κατάλογο με βασικούς δείκτες που θα είναι κύριοι άξονες για την αξιολόγηση της πολιτικής και την εφαρμογή του προγράμματος μεταξύ Περιφέρειας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός τώρα ο κατάλογος με τους βασικούς δείκτες και η επιλογή του προγράμματος θα πρέπει να συμφωνούνται κατά προτίμηση πριν το σχεδιασμό, πριν το προγραμματισμό. Βέβαια, από τη στιγμή που όλοι έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια, θα πρέπει ο κατάλογο τουλάχιστον των βασικών δικτών να κλείσει πριν τον ελιστικοποίηση του προγράμματο. Και να ξέρουμε ποιου βασικού δείκτε θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του προγράμματος, Βλέπουμε ότι η στοχοθέτηση εδώ σε ό,τι φορά τον αντίκτυπο του προγράμματος είναι ανεπαρκής. Είπε πριν από λίγο συνάδελφος ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ε, εκτός του προγράμματος που μπορεί να έχουν τεράστιο βάρος και σημασία σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση των αποτελεσμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του προγράμματος, σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από το περιεχόμενο του προγράμματος, πολύ περισσότερο από ό,τι από τους εξωτερικούς παράγοντες. Οπότε και το θέμα της αξιολόγησης ε, του input είναι σημαντικό, ε, αλλά και η αξιολόγηση του, το συνεπειών είναι σημαντική. Και δεν είναι άλλωστε δεδομένη, ούτε θα πρέπει να θεωρείται ως αυτονόητη για την περαιτέρω εκταμίευση των κονδυλίων. Κατά τη γνώμη μου και σε έναν ιδεώδη κόσμο, η πρώτη πιθανότητα για την εφαρμογή της στρατηγικής είναι τα κράτη-μέλη περιφερειες να συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους στόχους που επιδιώκει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη κατά προσέγγιση και το κόστος αυτού του προγράμματος και κατόπιν οι περιφέρειες στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν το πρόγραμμα υλοποιώντα τα αποτελέσματα και με βάση αυτά τα, αυτές τις επιδόσεις αυτό το βαθμό υλοποίησης να επιβραβεύονται με περαιτέρω δόσεις ε, για τη συνέχιση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος, ε, μάλλον υπάρχει πιθανότητα ακριβώς η περαιτέρω συνέχιση του προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα να είναι και λιγότερο δαπανηρή και πιο αξιόλογη Βέβαια, το κόστο που έχουμε δει σε προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού οφείλεται στο γεγονό ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων ε, και των, συγκεκριμένων στόχων θα είναι πιο δύσκολη για τι περιφέρειες. Και θα πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερη προσπάθεια στην εφαρμογή του προγράμματο για να επιδιώξει του στόχου, γιατί πλέον θα επήγεται να επιδιώξει του στόχου προκειμένου να λάβει τις, τα, τα επιπλέον κονδύλια. Νομίζω ότι όμω έτσι και οι δικαιούχοι και οι αρμόδιες αρχές θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για την καλύτερη επιδίωξη των αποτελεσμάτων και να είναι πιο αποδοτική στις εφαρμογές. Όλες αυτό είναι το ζητούμενο για όλους. Και πάλι όμως θα πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων προκαθορισμένη σαφή μεθοδολογία για να αποφασιστεί πότε ένα πρόγραμμα είναι επιτυχημένο ανάλογα με τους στόχους που πραγματοποίησε και σε περίπτωση που δεν υπήρχε πλήρης επιτυχία να υπάρχει και πάλι μεθοδολογία για το πώς θα δρομολογηθούν ανάλογα με την επιτυχία ή τα υπόλοιπα κονδύλια. Έχουμε, την τράπεζα, έχουμε εδώ την εμπειρία ε, και της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Μηχανισμού Γειτονίας. Οπότε μπορεί αυτές οι εμπειρίες να τις χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ουκρανία, Μολδαβία, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία είχαμε τέτοιες εμπειρίες, όχι μόνο από την Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή πιο μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τις γειτονικέ χώρες. Τώρα υπάρχει και δεύτερη εναλλακτική λύση, το Plan B, που θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Περισσότερα και απλούστερα κόστη». Βέβαια τώρα έχουμε κάποιες δαπάνες που εφαρμόζονται ε, με, διάφορο, με κυβερνόμενους βαθμούς επιτυχίες από διάφορες χώρες και ε, περιοχές. Και είναι και ανάλογα με το πώς γίνονται οι λογιστικοί υπολογισμοί και δεν αφορά τη διοικητικούς αρχή και το δικαιούχο απλώς αυτή η ανάλυση. Λοιπόν, τα αποτελέσματα όταν επιτευχθούν θα διευκολυνθεί η κατάσταση. Ήδη λοιπόν έχουμε αρκετή εμπειρία όσον αφορά το σχετικό θέμα και για να έρθω σε αυτό που είπα προηγούμενα, σε οριζόντιες πολιτικές που θα πρέπει να επιβάλλονται εκτός ε, συνοχής, του πλαισίου συνοχής, στους τομείς όπου είναι λογικότερο. Για να μην βαρύνεται η πολιτική συνοχής με αυτά τα άλλα ζητήματα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και τα προγράμματα CDE και F. Το F θα είναι υβρίδιο μεταξύ της παρούσης καταστάσεως και της προσέγγισης με στόχο τα αποτελέσματα. Δηλαδή θα προσπαθούμε για ελέγχου του κόστους και μετά θα επιβάλλουμε και άλλες απαιτήσει για τον έλεγχο των εκροών και των αποτελεσμάτων και να τιμωρήσουμε τους, τελευταίους, τους τελικούς δικαιούχους στις περιφέρειες που δεν πετυχαίνουν τα αποτελέσματα. Ένα τέτοιο ε, είδος ελέγχου ή κίνητρα ή κυρώσεις όσον αφορά την επιτύχηση των αποτελεσμάτων μπορούν να εφίστανται μόνο αν συμφωνούμε να μειώσουμε το βάρος των ελέγχων στην εισρωή και του, τον έλεγχο του κόστους προς τους δικαιούχους. Αν ισχύσει αυτό, θα τονίζαμε ότι μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να έχουν οι εκροές και τα αποτελέσματα. Και για να ολοκληρώσω, ερεσιμότητα είναι η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει, έχει συζητηθεί εκτεταμένα. Νομίζουμε ότι η αιρεσιμότητα έχει άμεση σχέση με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Τώρα, θα πρέπει να επισημοποιηθεί, η πλειοψηφία πάντως των χωρών μελών και των περιφερειών έχουν τέτοια εμπειρία από την αιρεσιμότητα. Και, είχαμε, και πριν χρησιμοποιήσουμε τον όρο αιρεσιμότητα προϋποθέσεις για τα προγράμματα που από τη στιγμή που αφορούν οι προποθέσει τα, τα αποτελέσματα, την αποδοτικότητα θα πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα και να θεσμοθετηθούν, να επισημοποιηθούν. Τώρα, εξωτερική αιρεσιμότητα και αιρεσιμότητα και σε σχέση με άλλε πολιτικές που έχουν κάποια σημεία επαφή με την πολιτική συνοχή δεν εμπίπτουν στο, στην εκτέλεση του προγράμματος και θα πρέπει καν να εξεταστούν εδώ. Και τέλος, ε, ε performance reserve, αποθεματικό αποδοτικότητας, δεν δικαιολογείται ούτε σε αυτή την περίοδο προγραμματισμού. Γιατί ούτε και το εθνικό αποθεματικό ήταν πολύ δημοφιλής λύση και γιατί αυτή την αποτυχημένη λύση να τη μεταφέρουμε και στην κοινότητα δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ και αφήνω λίγο χρόνο για τις συζητήσεις. Και ο τελευταίος μας ομιλητής θα μας μιλήσει από την εμπειρία που είχε από την επαρχία της Ουτρέχτης, ο κύριος Μπάρς Βαντεμπάρκ. Δεν μας έχει μείνει όμως πολύ χρόνος. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνει δυνατότητα να μιλήσω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το πιο σύντομος γίνεται. Πολλά υπόθηκαν ε, ήδη από τις προλαλήσαντες. I've been asked to uh, the requirements and διοικητικό δυναμικό και δυνατότητα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το σύστημα με έχει στόχο τη επιδόση, που δράστη επί των επιδόσεων και ποια είναι η προοπτική τη τοπική της τοπικής είναι οι, βασικοί μας όροι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική που εδράζεται από των αποτελεσμάτων. Τρία στάδια. Προτάσεις ευρωπαϊκή Επιτροπής. Σημαντική αρχή σύμπραξης εταιρικής σχέσεως και μετά δημιουργία δυναμικού. βλέπουμε κάποιες τάσεις στην ανάπτυξη πολιτικών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Κινούμεθα προς πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση εδαφική. Δημιουργούνται λειτουργικές περιφέρειες. Ο κ. Βανίστελ Ρόι γνωρίζει το παράδειγμα του στο Άιντχόβεν μάλλον. Το Άιντχόβεν που δημιουργήθηκε ένας πόλος προβληματισμού αν θέλετε. Συνεργάζονται διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης με κοινωνικούς εταίρους και αυξάνεται η τάση στην Ευρώπη. Και τομεακές πολιτικές ε, όλο και περισσότερο επιδιώκονται. Δημιουργούνται υπό στόχοι υποσύνολα στόχων που εξυπηρετούν, εξυπηρετούν τον γενικότερο στόχο όμως, τον ευρύτερο στόχο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λείπουν οι πόροι όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση συνδυάζει πόρους. Είδαμε οι Δήμοι του Βελγίου τι προβλήματα είχαν πρόσφατα με του προπολογισμού λόγω προβλημάτων της τραπέζης τέξια Και όλο και περισσότερο η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με εταίρους στον ε, τομέα τον ε, πολιτικών και των μη κυβερνικών οργανώσεων και δημιουργούνται διάφορες συνεργασίες. Πρέπει να υποστηριχθούν οι τοπικές αρχές για να εφαρμόζουν πιο ολοκληρωμένε πολιτικές σε εδαφικό επίπεδο. Εξωτές Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς έχουμε να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρώπη του 2020 να δίνει θεματικές προτεραιότητες. Ε, συμφωνούμε με αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πρέπει να είναι γενικότερο στόχο των συνθηκών αυτός και όχι μόνο για την Ευρώπη 2020. Θέλει θεματική προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα εγχειρίδιο στόχων θεματικών. Καλή ιδέα. Χρειάζεται όμω και ευελιξία για τι περιφέρειες να μπορούν να επιλέγουν τις πιο σχετικές για αυτές προτεραιότητες και δείκτες. Πρέπει να είναι προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω. Είμαστε αντίθετοι προς την ιδέα της Επιτροπής για στενή σύνδεση μεταξύ προτεραιότητας και κατηγοριών δαπανών και δικτών. Οι περιφέρειες πρέπει να είναι πλήρης εταίροι, να συμμετέχουν πλήρως στο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να γίνεται επιλογή στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και να λαμβάνεται υπόψη και στις ε, συμβάσεις σύμπραξης με τα κράτη-μέλη και στα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση στην Ευρώπη για προσεγγίσεις εκ των άνω προς τα κάτω όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στα κράτη-μέλη. Δεν αναμειγνύονται οι περιφέρειες και οι πόλεις στις επιλογές που γίνονται. Και αν θα επηρεάσουν και τη μελλοντική γενιά των εθνικών προγραμμάτων αυτές οι αποφάσεις, θα μην έχουμε εμείς έλλειψη ιδιοκτησία σε επίπεδο περιφερειακό. Και αν θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική συνοχή, αυτό το συνέστημα ιδιοκτησία, το ownership, είναι ένα από του βασικότερου όρου που πρέπει να πληρούνται. επιδόσεις Δεν γίνεται αυτό. Είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τα διάφορα προγράμματα σε τη σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Τα μικρά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε επίπεδο είναι μεγάλα τα με 15 κρατη μικρότερα με 12 κρατη Έχουμε πολλά προγράμματα σε πολλά επίπεδα. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα και τέσσερα περιφερειακά στην ε, Ολλανδία. Υπάρχουν προγράμματα στα κράτη-μέλη που βασίζονται επί πολλών ε, πόρων και ταμείων. Πώς να τα συγκρίνεις τα προγράμματα, είναι δύσκολο. Χρειάζεται καλή αξιολόγηση. Μετά, μια αξιολόγηση μετά από τρία χρόνια θα ήταν δυσκολότατη. Και να βραβεύεται το καλύτερο πρόγραμμα και τι καλύτερε επιδόσει, δεν νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο βάση ε, του ανταγωνισμού που μπορεί να γίνει και τη σύγκριση. Η αιρεσιμότητα αναφέρθηκε από τον ε, γείτονά μου. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπε. Η αιρεσιμότητα θα πρέπει να περιορίζεται στις επενδύσει τη πολιτική συνοχή. Ναι, στην εκ των προτέρων ερεσιμότητα και όχι στη μακροοικονομική ερεσιμότητα. Η ερεσιμότητα θα πρέπει να ταιριάζει με το περιφερειακό πλαίσιο και το εθνικό πλαίσιο και κάθε πόλη θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να επηρεάζει την συμμόρφωση με την ερεσιμότητα, τι διάφορε αιρεσιμότητε. Πρέπει να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση λοιπόν των εθνικών προγραμμάτων κλπ. Και, και στο σχεδιασμό και διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη των και την κατάρτιση συμβάσεων σύμπραξης για να υπάρχει πραγματική συνεργασία. Να αισθανόμαστε συμμετέχουμε και ότι είμαστε ιδιοκτήτε των προγραμμάτων και ότι κάνουμε τι σωστέ επιλογέ, ότι επιλέγουμε τι σωστέ προτεραιότητε, ότι επιλέγουμε του σωστού ε, δείκτε με του οποίου να συμμορφώνονται οι πόλει και οι περιφέρειε. Γιατί αυτοί στο κάτω-κάτω κάνουν τη δουλειά και θα πρέπει να συμμετέχουν και στι επιλογέ. Και φοβούμαστε ότι σε κάποια κράτη-μέλη ακολουθείται προσέγγιση που αφορά μόνο ε, συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κράτους μέλους. Για να πετύχουμε τη σωστή προσέγγιση με στόχο τα αποτελέσματα χρειαζόμαστε μια καλύτερη αρχή εταιρικής σχέσης, συνεργασίας. Αν θέλουμε να έχουμε καλύτερα προγράμματα, πιο εστιασμένα, σαφού, σαφείς στόχους εκ των προτέρων και εκπλήρωση της αρεσιμότητας. Όλοι οι φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι κοινωνικοί εταίροι και οι διάφορα ιδρύματα γνώσης σε όλες τις φάσεις των προγραμμάτων, προγραμματισμού και δεν χάρηκα ιδιαίτερος με τη διαφάνεια του γείτονα που εστιαζόταν μόνο στην εθνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μα, θα πρέπει να είναι διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα, με περισσότερε αρχέ δεσμευτικέ όσον αφορά τη σύμπραξη. Στον επόμενο κανονισμό πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστε προδιαγραφέ που καθορίζονται για την αρχή τη εταιρική σχέση για να γίνεται σεβαστό ο κανόνα, μάλλον ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση και πρέπει να είναι ευρεία η κάλυψη η χώρα μου αποτελεί την εξαίρεση σε πολλά κράτη-μέλη και στα νέα κράτη-μέλη δεν υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ε, διακυβέρνησης. Περιφέρειες, πόλεις ε, μένουν εκτός των διαπραγματεύσεων και του σχεδιασμό των προγραμμάτων. Απλώς εφαρμόζουν κάποια κομμάτια των προγραμμάτων. Και δεν μιλάμε έτσι για πραγματική διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων. Να πω κάτι για τη δημιουργία δυναμικού. Ξέρουμε ότι η έλλειψη διοικητικού δυναμικού εμποδίζει την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Είναι καλή ιδέα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημιουργία δυναμικού να μπαίνει στο θεματικό εγχειρίδιο, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Βασικό, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών και πόλεων σε πρόγραμμα όπως το Urban. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, διότι βλέπω κάποια κόπωση στα παλαιότερα κράτη-μέλη. Δεν θέλουν να συνεχίσουν πολύ τη διασύνδεσή τους με τις περιφέρειες και τις πόλεις των νέων κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν οι πόλεις και οι περιφέρειες θα πρέπει να παρακινηθούν για να, των παλιών κρατών μελών συνεργαστούν με, κρα, με πόλεις και περιφέρειες των νέων κρατών μελών και η επιβολή, η εφαρμογή της αρχής εταιρικής σχέσης χρειάζεται μεγαλύτερο δυναμικό περιφερειακό σε επίπεδο για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αν θέλετε καλύτερες πολιτικές με βάση που θα έχουν σαν στόχο καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να υπάρχουν σαφείς δείκτες, σαφείς στόχοι και εκ των προτέρων αρισιμότητα, αλλά και επαρκής ευελιξία για την τοπική αυτοδιοίκηση να εφαρμόζει πραγματικά ολοκληρωμένη εδαφική πολιτική. Αν η πολιτική συνοχή είναι κάτι παραπάνω από του στόχου Ευρώπη Ευρώπη 2020, θα θέλουμε κάτι τέτοιο και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα τη πολιτική συνοχή, τότε χρειαζόμαστε πραγματική δικυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα, ξεκινώντα από το σχεδιασμό των εθνικών ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Χρειάζεται απλούστευση των κανονισμών, αλλά όχι μόνο το γενικό των γενικών πλησίων πρέπει να αλλάξει, ε, συζητείται και η αλλαγή της οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες. Πρέπει σίγουρα να ακουστευτεί και αυτό. Υπογραμμίζω τη σημασία της διακυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα. Ε, πες μου και θα, τέλος πάντων, πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Κυρίες και κύριοι, ε, ακούσαμε τις διάφορες παρουσιάσεις. Έχετε τα πάντα επί χάρτου. Σημαντικό αυτό. Για να συμμετέχουν όλοι. Πρέπει να τελειώσουμε μάλλον σε πέντε λεπτά. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα λεπτό. Θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και αν είναι σαφείς ε, και σύντομες μπορεί να προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Αλλά Τώρα βρισκόμαστε στα μέσα της διαδικασίας προετοιμασίας της επόμενης περίοδου. Οπότε, αν απευθύνουμε άμεσα προς συγκεκριμένους ομιλητές της ερωτήσεις μας, μπορούμε να λάβουμε και διμερώς απαντήσεις. Ας ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις. Είδα ότι η κυρία Μπρίζο Μπόχατα ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο κυρία Μπερζομπόχατα. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που εγκαινιάσαμε τη συζήτηση αυτή, γιατί έχω την αίσθηση ότι όταν λέω ότι θα πρέπει να πιάνω τόπο τα λεφτά, είναι σαν να μιλάμε μόνο για λογιστικά και διοίκηση. Αυτή την εντύπωση δίνουμε μερικές φορές λέμε να αποφύγουμε τα σφάλματα, τις παρατυπίες, να έχουμε χαμηλό επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, αλλά πολύ σπάνια μιλούμε για την αξιοποίηση των κονδύλιων, για την αποτελεσματική τους χρήση. Πρέπει περισσότερο να προσανατολισόμαστε προς αυτό το στόχο, τα αποτελέσματα μιλήσαμε για πολλούς και διάφορους στόχους καταμέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Στους Δήμους όμως και τις κοινότητες έχουμε πρόβλημα με την καταμέτρηση και την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Σε ορισμένα προγράμματα είναι εύκολο να ποσοτικοποιήσουμε τα αποτελέσματα ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων ή να μετρούμε ένα μονάδα. Αλλά πώς θα αποτιμήσουμε την ικανοποίηση, για παράδειγμα, των κατοίκων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο θα μας πει ο Δήμος δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε την ικανοποίηση, άρα δεν μας ενδιαφέρει το αρνητικό αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει και ένα άλλο άκρο. Όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε μαθηματικές μεθόδους στην καταμέτρηση της ικανοποίησης από ένα πρόγραμμα. Χαίρομαι λοιπόν που εκπρόσωποι του, του ακαδημαϊκού κόσμου μίλησαν για απλές μεθόδους Εύχριστε που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν ακόμη και σε μικρές κοινότητε. Και δεν μιλάω για τι μακροπεριφέρειες, γιατί οι πιο μεγάλες περιφέρειες ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και πιο εκλεπτισμένε και εξαζητημένες μεθόδους. Αλλά θα πρέπει να έχουμε απλές μεθόδους να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και η μικρή κοινότητα. Και φυσικά να είναι εύχριστε και για τους ανθρώπους που θα προετοιμάσουν και θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Θα μπορούσαμε επίσης ε, να βελτιώσουμε την επιμόρφωση των αρμοδίων των κοινοτήτων, ώστε να εφαρμόζουν αντίστοιχες με μεθοδολογίες και στις καθημερινές τους δραστηριότητες και εργασίες. Δεν έχω λοιπόν τόσο ερώτηση όσο να ζητήσω από τους εκπροσώπους ε, του ακαδημαϊκού κόσμου να επεξεργαστούν τέτοιες μεθόδους απλές και εύχριστες. Γιατί υπάρχουν στον επιχειρηματικό κλάδο, αλλά δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε πολλές φορές. Σύντομες απαντήσεις. Ο Γιάννη είναι πρωταθλητής στις ε, σύντομες ε, συνοπτικές και εύστοχες ερωτήσεις. Α, αυτή τη φορά όχι όμως, λέει ο κύριος Όλμπριχτ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις κι εγώ, γιατί δεν ήμουν παρόν καθόλου τη διάρκεια της ακρόαση, Παρατήρηση πρώτη. Όντως δεν διαλέξαμε καλά την ώρα για την ακρόαση αυτή, γιατί ήμασταν τρεις και ο Κούκος. Μείναμε ελάχιστοι μετά την δύσκολη αυτή ψηφοφορία. Και όσοι παρακολούθησαν την ψηφοφορία μετά έφυγαν. Ενώ το θέμα είναι και πολύ σημαντικό και επίγον. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση άλλη φορά γιατί το θέμα της αποτελεσματικότητας, καταμέτρησης των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης είναι από τα πιο καθόδη ζητήματα και τα πιο δύσκολα. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένο και είπαμε ότι θα έχουμε μια πολιτική που θα προσανατολίσει στα αποτελέσματα. Ε, μα όλες οι πολιτικές δεν προσανατολίζονται στην υλοποίηση ενός των αποτελεσμάτων. Αλλή μόνο λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε πολιτικέ στην Ευρώπη που θα, θα προσανατολίζονται στα αποτελέσματα. Δηλαδή, μέχρι τώρα οι πολιτικέ μα δεν είχαν στόχο να υλοποιήσουν αποτελέσματα. μόνο. Φυσικά θέλουμε πολιτικές πιο αποτελεσματικές, αλλά όχι ότι μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές, απλώς θέλουμε να βελτιώσουμε αυτή την αποτελεσματικότητα. Έχουμε και το θέμα της συζήτησης απαλλαγής. Έρχεται στη συζήτηση της απαλλαγής στο ελεκτικό συνέδριο και το ελεκτικό συνέδριο δεν ασχολείται με τις πολιτικές που στηρίζονται σε αποτελέσματα, αλλά με τις πολιτικές που στηρίζονται σε σωστά λογιστικά στοιχεία. Και δεν φταίει γι' αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό είναι ζήτημα διοίκηση. Η διοίκηση πρέπει να ελέγχει και τα λογιστικά, τα έγγραφα. Και μιλούμε για το επίπεδο, κινδύ... επίπεδο ελέγχου, όχι ε, επίπεδο λάθους, συγγνώμη, σφάλματος, όχι στα αποτελέσματα, αλλά στις διαδικασίες. Και ζητά το ελεκτικό συνέδριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πιο αυστηρό έλεγχο για να μειωθούν τα σφάλματα, το ποσοστό σφάλματο. Ποιο όμω θα είναι το κόστο του ελέγχου που θέλουμε για να αποφύγουμε τα σφάλματα. Γιατί αν ο έλεγχο είναι αυστηρότερο, τότε θα μειωθεί η προσπάθεια που αφιερώνουμε στα αποτελέσματα. Και τα σφάλματα στην πολιτική συνοχής οφείλονται εν μέρη στι διαδικασίε δημοσίων συμβάσεων, που είναι πολύ διαφορετικέ στι χώρε μέλη. Και υπάρχει το θέμα τη επιλεξιμότητα. Εσεί μιλήσατε κάποια στιγμή για τι δημόσιε συμβάσει. Στο Κοινοβούλιο την ίδια στιγμή η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς εξετάζει το θέμα των δημοσίων συμβάσεων και της σχετικής οδηγίας. Εμεί στη δική μα Επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξη σχεδόν κανένα δεν ξέρει ότι στο, δημόσιο, στο δημοσιονομικό κανονισμό υπάρχει ένα ε, εκτενές κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Έχουμε λοιπόν και τον κανονισμό που έχει ένα κεφάλαιο για αυτό το θέμα και την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Και τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε αντιφατικά αποτελέσματα και να δημιουργηθεί σύγχυση. Γιατί και μέσα στο ίδιο το Κοινοβούλιο έχουμε δύο διαφορετικά όργανα για το ίδιο θέμα. Χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό λοιπόν. Επίσης, μιλήσαμε για το ζήτημα των δικτών. Ταυτόχρονα αναφερθήκαμε και στο αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Λυπούμαστε, αλλά η διερμηνία σταματάει αυτή τη στιγμή. Καλώς σας μεσημέρι. But not what about the evaluation, but what about the follow-up of evaluation? Because this is the question. If we have the much more developed procedures on evaluation, we should have some kind of follow-up Because if we follow up, this is just the exercise. Very interesting. Very interesting for the scientists. Uh, το πρόβλημα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε την παρακολούθηση της αξιολόγησης ε, και ενώ θα συνεχίσουμε την αξιολόγηση για το πρόγραμμα που τελειώνει, να διασφαλίσουμε και τη συνέχεια για το επόμενο πρόγραμμα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αλλιώς θα συζητούμε συνέχεια ε, πολιτικές που προσανατολίζονται στα αποτελέσματα, ενώ οι μακροοικονομίες εξετάζουν ακόμη την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, λέει ο μιλητής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τώρα τη συζήτηση και όντω αυτή τη στιγμή σταματάει και η διερμηνία γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ το ωράριο εργασία. Καλό σας μεσημέρι.